Bien, Σας προτείνω να ξεκινήσουμε κύριε Πρόεδρε. Πρώτο σημείο. Είδατε νομίζω την ημερήσια διάταξη. Γύρω από την ημερήσια αυτή διάταξη και σύμφωνα με αυτά που περιλαμβάνονται στο Κόμπου News, το σημείο 4 που αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό του 13 αναβάλλεται και θα συζητηθεί την ημέρα Πέμπτη. Γιατί αυτή την εβδομάδα συνεδριάζουμε με κάπως περίεργο τρόπο θα έλεγα, ευτυχώς. Οι δύο μισές μας μέρες είναι σήμερα το απόγευμα και θα ξαναβρεθούμε την Πέμπτη όπου θα υπάρξει στις δύο συνάντηση των συντονιστών και η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα συνεδριάσει από τις 3 ε, μέχρι τις 6.30 αλλά σε διαφορετική αίθουσα θα είμαστε στον έκτο όροφο του κτηρίου Αντάλλα. Σήμερα το απόγευμα θα ψηφίσουμε γύρω στις 5 και θα τελειώσουμε τη συνεδρίαση στις 6 το απόγευμα προσκαλώντας τους συναδέλφους της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών όπως επίσης και το συνεισηγητή τους, τον κύριο Ριβελίνη, για να συζητήσουν με την κυρία Γκρέσλε και να μας παρουσιάσουν τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό κανονισμό. Στρέφομαι προς τον κύριο Φέρνο. Ο κύριος Φέρμ πήρε μέρος σε ένα τρίλογο με το Συμβούλιο για τα project bonds. Κύριε Φέρμα, θέλετε να μας κάνετε μία παρουσίαση ή θέλετε να κάνετε μια παρουσιαση θελετε να αναφορά, τι ακριβώς. Νομίζω ότι μπορώ να σας κάνω την παρουσίαση πάρα πολύ σύντομα. Ήταν η πρώτη συνάντηση του τριμερούς διαλόγου, ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Είχαμε αρκετά θέματα τα οποία ήταν πολύ δύσκολα θα έλεγα, θα μπορούσαν να είναι τουλάχιστον πολύ δύσκολα το Συμβούλιο θέλει μια στρατηγική εξόδου από τα project bonds πριν καν ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την έκδοσή τους. Αυτό σημαίνει ότι προβλέπουν την αποτυχία αυτών των ομολόγων. Προφανώς είναι μια πιλωτική φάση. Είναι σαφές ότι αν τυχόν τα πράγματα πάνε καλά θα μονιμοποιηθούν. Αν δεν πάνε καλά θα διακοπούν. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι εξ αρχής να βρούμε έναν τρόπο εξόδου, έτσι θέλει το Συμβούλιο, Κάτι τέτοιο θα καταστήσει, θα έλεγα, στις χρηματαγορές το πρόγραμμα αυτό λιγότερο αξιόπιστο. Πιστεύαμε ότι το Συμβούλιο θα είναι άγριο σε σχέση με το πρόβλημα, αλλά δεν ήταν και τόσο. Είπαν ότι θα προσπαθήσουν να βρουν μια νέα διατύπωση αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επανέλθουν στο Κορεπέρ για να πάρουν μια νέα εντολή για την αλλαγή αυτή και αυτό δημιουργεί ένα χρονισμού πρόβλημα. Πάντως ελπίζω να πετύχουμε τον στόχο που έχουμε να ψηφίσουμε την πρώτη ανάγνωση, δηλαδή την 1η Μαΐου. Πάντως, 21 Μαΐου συγγνώμη. Δεν ενδιαφέρονται ακριβώς για όλες τις πολιτικές απόψεις τις οποίες είχαμε εμείς, όπως επίσης και για τις επιλογές για ένα πρόγραμμα θα έλεγα πιο φιλόδοξο έκδοσης ομολόγων, σαν παράδειγμα εισαγωγή δυνατοτήτων έκδοσης ομολόγων σε τομείς όπως η αηφορία, το περιβάλλον κτλ. Όχι, πάντως αυτό δεν είναι σοβαρό πρόβλημα, είναι πρόβλημα ορολογίας περισσότερο. Πάντως η αναφορά που σας κάνω συνολικά πρέπει να χαρακτηριστεί θετική και νομίζω ότι έχουμε μια αρκετά σοβαρή δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια απόφαση την 21η του μηνός Μαΐου. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Λαμασούρ, ευχαριστώ κύριε Φέρνα. Την προηγούμενη Κυριακή ξέρετε ότι έγιναν εκλογές προεδρικές στη Γαλλία. Πάνω σε αυτό... Je dis bien sur ce sujet précis, parce que notre séance est publique, il faudrait pas y malentendu sur mes propos. Sur ce sujet... Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, λέει μετά από μια τεχνική διακοπή ο Πρόεδρος, θα πρέπει να υπάρξει μια θετική, θα έλεγα, ε, έκβαση από πλευράς της γαλλικής πλευράς, από πλευράς γαλλικής. Για το θέμα δηλαδή των ομολόγων, των ευρωομολόγων ή προγραμματικών ομολόγων όπως θέλετε, ε, θα υπάρξει θετική άποψη της Γαλλίας, είναι σαφές. Μιας και τώρα βρισκόμαστε στο φάση των ανακοινώσεων, θα πρέπει ναι. να σας πληροφορήσω ότι αντιμετωπίζουμε ορισμένες δυσκολίες και αυτό δεν θα σας εκπλήξει. Να πείσουμε τα άλλα δύο όργανα και ιδιαίτερα το Συμβούλιο να φέρει εις πέρας στο Συμβούλιο την κοινή ανάλυση που είχαμε ξεκινήσει για την κατανάλωση των πιστώσεων πληρωμών και για την δυνατότητα, θα έλεγα, ε, εξασθένησης των ΡΑΛ. Κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου, που ήταν ο πρώτος τριμερής διάλογος, ο οποίος είχε αποκλειστικά, θα έλεγα, σαν στόχο μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τον προϋπολογισμό του 2013, η Προεδρία της Δανίας είχε δεχθεί την πρότασή μας για μια κοινή συνάντηση των τριών ε, οργάνων γύρω από το θέμα αυτό. Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν την οποία είχα κάνει εξ ονόματος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου μετά από αίτημα των μελών του Κοινοβουλίου στην διαβούλευση στο τέλος του προηγούμενου χρόνου για τον προϋπολογισμό, των προσχέδιο του 2013, λόγω της αβεβαιότητας που είχε δημιουργηθεί στην τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης για το ακριβές ύψος των αναγκών στις πιστώσεις πληρωμών για το 2011. Ήδη λοιπόν από τις αρχές του 2012 εμείς μείναμε σε μια κάποια φάση αβεβαιότητα σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες των πιστώσεων πληρωμών. Η συνάντηση αυτή λοιπόν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη. Δυστυχώς η Προεδρία της Δανίας εκπροσωπήθηκε στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου από τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είναι προφανώς υπεύθυνος για θέματα καθαρά προϋπολογισμού, δεν επιβεβαίωσε την συμφωνία αυτή της Προεδρίας και μάλιστα ανέφερε ότι στα πλαίσια της συνάντησης δεν ne souhaitait pas s'exprimer en tant que tel et Πάλι έχουμε μια τεχνική διακοπή, συγγνώμη δεν θα υπάρξει εκπροσώπηση σε πολιτικό επίπεδο της Προεδρίας αλλά σε επίπεδο τεχνοκρατών. Υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό με την διερμηνία, διακόπτεται η... Pour la langue tchèque, pour le polonais, pour le hongrois. Alors, quel est, quel est le problème Il n'y a aucune traduction Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τη διευμηνία. Υπάρχει μια διακοπή μετάδοσης. My voice is disappearing. Πώς δεν ακούγεται η φωνή μου όλο και λιγότερο. Άμα ακούτε μία λέξη στις δύο μπορεί να αρκεί, δεν πειράζει ίσως. Τα μισά να ακούτε. Μήπως οι τεχνικοί ξέρουν Πώς διορθώθηκε λέει. Διορθώθηκε τσεχικά, ουγγρικά, πολωνικά διορθώθηκε, διορθώθηκε και πολωνικά. Και ιταλικά, ναι. Συνοψίζω. Η ιδανική προεδρία υπαναχώρησε. Εδώ μεταξύ με τους συντονιστές είχαμε πει να οργανώσουμε δύο συνεδριάσεις, μία πρώτη τεχνικού επίπεδου και μία δεύτερη πολιτικού επίπεδου με τους αρχηγούς των αντιπροσωπιών για τα τρία όργανα. Λόγω όμως της θέσης της Δανικής Προεδρίας και σε συμφωνία με τους συντονιστές και συντονίστριες αποφασίσαμε τα εξή. Αύριο 9 Μαΐου θα γίνει μια συνάντηση τιμερής μεταξύ των εισηγητών μας και της Κομισιόν που είναι εδώ παρόν, παρούσα. Όταν λέω εισηγητές και εισηγήτριες εννοώ ότι μπορούν και τα ενδιαφερόμενα μέλη, ιδίως οι σκιώδεις, να προσέλθουν. Δημερίς, λοιπόν. Και εκεί ελπίζουμε να υπάρξει κάποια πρόοδος μεταξύ κομπούς και κομισιών έτσι ώστε στις 30 Μαΐου να μπορέσει να οργανωθεί συνάντηση, συνεδρίαση με σε μένα, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και με επικεφαλή τον κύριο Λεβαντόφσκι από την άλλη μεριά. Ούτως ή άλλως πάντως το Συμβούλιο δύσκολα θα μπορέσει να απουσιάσει τελείως. Αν δεν θέλει να εκφραστεί, δεν θα εκφραστεί βέβαια, αλλά Νομίζουμε ότι για αυτό το πολύ τεχνικό θέμα και τεραστίω πολιτικό, ιδιαίτερα στους καιρούς που ζούμε, θα έχουμε τουλάχιστον την εγγύηση ότι υπάρχει μια συμφωνία, ότι θα υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιών όχι για τα ποσά τα ίδια, αυτό είναι θέμα της διαπραγμάτευσης, αλλά για τον τρόπο υπολογισμού των αναγκών και καθορισμού των επιλογών για να μειωθούν τα ράου. Έτσι θα διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση για τον προπολογισμό του 12. Να, αυτά ήθελα να σας πω. Και επειδή αύριο θα γίνει αυτή η λεγόμενη τεχνική συνάντηση, τεχνική τη λέμε, αλλά αφού έχουμε όλους μας τους συζητητές και συζητήτρες, ήδη από την Πέμπτη θα μάθουμε τι συμβαίνει. Αυτά λοιπόν κατά τα άλλα. Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι γραμμένες εδώ στα νέα της κομπούς και εκτός αν ακουστούν αντιρρήσεις εγκρίνουμε τα πρακτικά της 29ης Μαρτίου. Τώρα. Τώρα... Επειδή το 4 έχει αναβληθεί για μεθαύριο ή για αύριο, περνάμε στο 5. Το σχέδιο διορθωτικού προλογισμού αριθμό 2 του 2012, Ταμείο Αλληλεγγύης για τις πλημμύρες στην Ιταλία. Η συγγήτρια μας Φραγκίσκη έχει το λόγο, Μπαλτζάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη είχαμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προηγούμενες συναντήσεις μας. Έχουμε κάτι το καινοτόμο τώρα, μια επιστολή του κυρίου Λεβαντόφσκη, του Επιτρόπου, και αναδιατυπώνει την πρότασή του σχετικά με την κάλυψη του προβλήματος των πληρωμών. Γνωρίζετε ότι το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η έλλειψη 18 εκατομμυρίων που ζητήθηκαν έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα τα ποσά για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Η πρόταση η πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μια αναθεώρηση των μέγιστων ποσών που ήταν διαθέσιμα για πέρυσι ε, είναι μια πρόταση του κυρίου Λεβαντόσκη ε, για την οποία θα αποφασίσει το Συμβούλιο σύντομα. Υπάρχει όμως και το θέμα των επιστροφών εδώ. Ο κύριος Λεβαντοσκη προσπαθώντας πάντα να συγκεντρώνει την προσοχή μας στο θέμα των πληρωμών που όπως γνωρίζετε είναι ένα από τα πιο περίπλοκα και συζητημένα θέματα για τον προϋπολογισμό φέτος προτείνει να επαληθεύσουμε προσεκτικά το επίπεδο εφαρμογής του πακέτου των προγραμμάτων, ιδιαίτερα τα προγράμματα της ενέργειας που συνδέονται με το οικονομικό πρόγραμμα ανάκαμψης και προτείνει ένα πακέτο 350 εκατομμύρια μέσα στο οποίο υπάρχουν προβλέψεις για υποχρησιμοποίηση λόγω ακριβώς του περίπλοκου χαρακτήρα και της αργής ταχύτητας αυτού, αυτών των προγραμμάτων. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν ανάκαμψης είναι περίπλοκα και γι' αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν περισσέψει σε εισαγωγικά 350 εκατομμύρια και προτείνει ο Επίτροπος να τα χρησιμοποιήσουμε για τις βέβαιες ανάγκες, δηλαδή τα 18 εκατομμύρια του Ταμείου Αλληλεγγύης και για τη χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων έρευνας τα οποία πάρα πολύ σύντομα μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ανάγκη από άμεσες πληρωμές. Συνεπώς λοιπόν η πρόταση του Επιτροπή τρόπου Λεβαντόφσκι είναι από τη μία να, σε επίπεδο πολιτικό να υπάρχει πάντα συζήτηση για το θέμα των πληρωμών γιατί το πρόβλημα μέχρι το τέλος του χρόνου ε, θα χειροτερεύσει θα έλεγα, το θέμα των πληρωμών θα χειροτερεύσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και είναι απαραίτητο να γίνει μια σωστή αναθεώρηση του προγράμματος έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν και χρήματα από το πρώτο πακέτο των επιστροφών είτε για το Ταμείο Αλληλεγγύης είτε για τα προγράμματα τα, για τα οποία θα χρειαστεί να δώσουμε χρήματα πριν το τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Μπαλθάνη. Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι μάλλον βρήκαμε ένα νέο κοίτασμα ρευστότητας εφόσον συμφωνήσουμε, που θα επιτρέψει τουλάχιστον να χρηματοδοτήσουμε ε, το Ταμείο Αλληλεγγύης για τη Λιγουρία και την Τοσκάνη. Ταυτόχρονα, τα κακά είναι ότι αυτό η ακριβώς η δυνατότητα δείχνει ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα των πιστώσεων οι οποίες είχαν προβλεφθεί ως προερχόμενες από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ανάκαμψης από την οικονομική χρήση δεν χρησιμοποιήθηκαν. Οφείλουμε λοιπόν να βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα για αυτού του τύπου τις αποφάσεις, για αυτού του τύπου τις διαδικασίας και σε επίπεδο δημοσιονομικού κανονισμού και σε επίπεδο βέβαια πολιτικών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στα πλαίσια του προγράμματος ανάκαμψης. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Υπενθυμίζω εδώ ότι υπό την αίρεση βεβαίως του χρονοδιαγράμματος υιοθέτησης της θέσης του Συμβουλίου η προθεσμία για τις τροπολογίες, εφόσον υπάρχουν τροπολογίες, θα καθοριστεί για την 24η Μαΐου. Λοιπόν, δεν σας δημιουργεί πρόβλημα η ημερομηνία, ε, κυρία εισηγήτρια ανάλογα πάντα και με το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου. Αυτά τελειώσαμε με το 5, περνάμε τώρα στο 6 παρακαλώ. Έχουμε εδώ να κάνουμε με την έκθεση του κυρίου Φρανσουά Αλφονσί, ο οποίος έχει να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του για την κοινή αλλιευτική πολιτική. Και προτείνει τώρα πλέον μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Αλφονσί έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Donc, euh, nous sommes sollicités pour un avis. Γνωμοδότηση είναι αυτή για την κοινή αλληλευτική πολιτική από το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει να βρει ένα δρόμο για να φτάσει σε μια απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε ένα πόρο που είναι υπό εξαφάνιση, υπό απειλή, αλλά και μια οικονομική δραστηριότητα για να μπορέσει η Ευρώπη να ασκεί αυτή την αληφτική δραστηριότητα. Το 2009 εξετάστηκε μια πράσινη βίβλος για την αναθεώρηση τη κοινή αληφτική πολιτική και κατέληξε ότι δεν είχαν τελειώσει ακόμα τα βάσανά μα και δεν είχαμε ακόμα αληφτική πολιτική στην Ευρώπη που να ε, είναι συμβατή με τη διαφύλαξη και την ανανέωση των ειδών γιατί ήταν πολύ μεγάλη υπεραλίευση την προηγούμενη περίοδο. Από εκεί και πέρα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα και να ορίσουμε κάποιες προτεραιότητες. Δηλαδή, να λαμβάνουμε καλύτερα υπόψη το θέμα της περιβαλλοντικής αηφορίας και βιωσιμότητας. Επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλες οι απορρίψεις κάποιων ειδών ε, που αλλιεύονται και τελικά ξαναρίχτονται στη θάλασσα και το θέμα της υπερβολικής χωρητικότητας του στόλου μας, του αλευτικού που για την Ένωση είναι και κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα πάρα πολύ οξύ και ανισχυτικό. Τώρα, τι μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικώ. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά στα πλαίσια ενός ταμείου το οποίο εάν τελικά ε, περάσουν είναι 6,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Μικρή μείωση, αλλά είναι της τάξης του περασμένου μεγέθους. Και στόχο έχουν αυτά τα κονδύλια να προωθήσουν μια σειρά προσανατολισμών μέτρων, δηλαδή να μειωθούν και να ε, σταματήσουν οι ε, απορρίψεις, η υπεραλίευση κάποιων ειδών, ε, να μεταβάζονται οι άδειε ε, και υπάρχουν πάντα κάποιες ε, αμφισβητήσεις λόγω επιστημονικών δεδομένων, δεν συμφωνούν μεταξύ τους τα στοιχεία. Θα μπορούσα να σας κάνω μια λεπτομερή αναφορά για το κανονισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παράκτελεια για το σύστημα της μεταφορές εκχώρησης αδειών ε, τελικά θα καταλήξει στον αφανισμό ε, ενός ολόκληρου επαγγελματικού κλάδου που είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ζωής στις τοπικές παράκτιες κοινότητες. Και ε, στη διαχείριση των ακτών συμμετέχουν αυτοί οι πληθυσμοί, θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθούν. Επίσης είναι και το θέμα της Natura 2000 που θα πρέπει ε, να ε, εφαρμοστεί σε όλες τις θάλασσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί προσανατολισμοί συνεπώς είναι καλοί και μπορούμε να δώσουμε ευνοϊκή ε, γνωμοδότηση. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε, ο Γιώραν Φέρμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομο σχόλιο εξ ονόματος της κυρίας Τρελιέ που συνεχίζει ακόμα την προεκλογική εκστρατεία στη Γαλλία. Τη μετεκλογική, αλλά όχι έχουν και άλλες εκλογές όπως γνωρίζετε. Θα ναι. ήθελα να πω δύο λόγια. Συμφωνεί γενικά ε, με τον κύριο Αλφονσί. Ε, θα πρέπει η γνωμοδότησή μας να είναι σύντομη. Θα επανέλθουμε σε άλλα σημεία της νομοθετικής ε, πρότασης για την Αλία εν ευθέτω χρόνο. Θέλει εκείνη να τονίσει ιδιαίτερα ότι είναι δημόσιο αγαθό η αλληλευτικοί πόροι και θα πρέπει να τους προστατεύουμε όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για την παγκόσμια επιστηστική ασφάλεια. Επίσης δεν είναι μόνο η αλληλεία, η δατοκαλλιέργεια και λοιπά, πολύ σημαντική για συγκεκριμένες παράκτης περιοχές και εδώ θα χρειαστεί να υποστηριχθούν και στο μέλλον. Είναι σαφές ότι υποστηρίζουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική που έχει ως στόχο την αηφόρο αλληλεία με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει οικονομικά να είναι βιώσιμη για τις αλληλευτικές κοινότητες που εξαρτώνται από τη δραστηριότητα αυτή και στο μέλλον. Αυτό τι σημαίνει. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι ανάγκες χρηματοδότησης για αποτελεσματική διαχείριση των αλλιευτικών πόρων και σίγουρα εδώ θα χρειαστούν περισσότερες επιστημονικές έρευνες κτλ. Και αν χρειαστεί να βελτιωθεί η δραστηριότητά μας, να αλλάξουν ε, τα αλλιευτικά σκάφη, πηγαίνουμε προς μια πιο επιλεκτική αλλιευτική πολιτική και θα πρέπει να βελτιωθεί ε, ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται τα βιολογικά στοιχεία. Θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε τα στοιχεία. Θα βασιστούμε βέβαια εμείς για τη γνωμοδότηση στην έκθεση της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Έχουμε νέα προαπαιτούμενα για την ελευτική πολιτική για να γίνει αυτή βιώσιμη. Και θα πρέπει να δούμε πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν εντός των ορίων και των ορφών που είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε. Θα επανέλθουμε Όλα αυτά τα λέει η κυρία Γκριλιέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ο Καρλ Χάγκλουντ. Ευχαριστώ. Σύντομα. Είναι πολύ εύκολο να συμφωνήσει κανείς με τα όσα προτείνει ο Φρανσουά. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας όταν ε, άρχισε την μεταρρύθμιση, την προσπάθεια της Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι θα πρέπει να είναι ριζική αυτή η μεταρρύθμιση και πολύ σοβαρά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πολύ σπάνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημόσια δηλώνει ότι έχει αποτύχει σε μια πολιτική της και χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση. Δεν συμβαίνει αυτό κάθε μέρα. Και τα περισσότερα αλλιεύματα, τα περισσότερα είδη στην Ευρώπη υπεραλλιεύονται. Και αν δεν το αλλάξουμε, θα απειληθεί πραγματικά ο κόσμος που εξαρτάται από την αλία, όπως είπε ο Γιώργος. Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσεις εισόδημα και επιβίωση αυτού του κλάδου είναι να είναι μια σωστή ε, και οικολογική προσέγγιση για τον αριθμό των αλιευμάτων. Αν έχουμε αηφόρο προσέγγιση στο τεινικές θα αυξηθεί και το ε, εισόδημα. Αλλά αυτή τη στιγμή και βραχυπρόθεσμα πρέπει να ε, μειωθεί η αλληλευτική δραστηριότητα. Είναι σημαντική αυτή η φάση, ε, η πρώτη φάση που θα μειωθεί η προσπάθεια και θα πρέπει να το συζητήσουμε κι εμείς. Έχω τη χαρά να είμαι ένας από τους ηγητές για τη μεταρρύθμιση και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αλίας. Ασχολούμαι πολύ εντατικά με αυτά τα πράγματα. Είναι όντως πρόκληση, αλλά υπάρχουν δυνατότητες και πολιτικές, ήδη από τη σημερινή ελευτική πολιτική, που θα μπορούσαν, πώς να το πω, να χρησιμοποιηθούν αλλιώς, ειδικά η χρηματοδότηση. Με άλλα λόγια, δεν είμαι πεπισμένο ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για την κοινή αλληλευτική πολιτική, αλλά μπορούμε να τα δαπανίσουμε καλύτερα για να ξεπεράσουμε αυτή τη φάση και να προχωρήσουμε σε μια πιο βιώσιμη αλλήλεια. Και είμαι βέβαιο ότι συμφωνούμε με τον εισηγητή και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία για να εκφραστεί με τρόπο στεναρό και η φωνή τη Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Σα κάτι ευχαριστώ. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, για ένα τέτοιο θέμα είναι σημαντική η γνωμοδότησή μας. Τα ποσά που συζητάμε είναι σημαντικά, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Διαπιστώσαμε, γιατί και εγώ κλαίγομαι σε μια περιοχή νοτιοδυτικά της, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της Ατλαντικής ακτής και της Μεσογειακής Τιάφτης ως προς την αλληλεία. Όπως και άλλοι διαπίστωσα και εγώ λοιπόν ότι στο παρελθόν οι κοινοτικές επιχορηγήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την καταστροφή ή η καταργηση πλοιαρίων για να μειωθούν οι αλλιεύσεις και ταυτόχρονα ενεθάρινε την αγορά πιο σύγχρονων αλλιευτικών πλοιαρίων για μεγαλύτερη ασφάλεια μεταξύ άλλων των πληρωμάτων λιγότερα δηλαδή πλοιάρια αλλά που αλλιεύουν περισσότερο και υπάρχουν πολλά είδη που αυτή τη στιγμή απειλούνται από την υπεραλία αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός ούτε και των αλλιέων γι' αυτό η Κομισιόν έκανε πολύ καινοτόμες προτάσεις και κατανοώ γιατί οι Υπουργοί Αλλιείας σε πρώτη, η πρώτη τους αντίδραση ήταν πολύ μέτρια. Κοντά στην Ένωση, μια φορά και μέσα της, υπάρχουν χώρες που κατάφεραν να εφαρμόσουν μέτρα που έδιναν, αύξαναν την ευθύνη των αλλιέων και διασφάλιζαν και την ανανέωση του πόρου των αλλιευμάτων δηλαδή. Αυτό βέβαια έγινε κυρίως σε μικρών διαστάσεων εκμεταλλεύσει. Υπάρχουν λοιπόν επαναλαμβάνω μέρη όπου τα κατάφεραν να το πετύχουν αυτό. Η Κομισιόν δεν έχει ως καθήκον να μας πει ποια είναι η καλύτερη μέθοδος, αυτό είναι θέμα των εισηγητών μας, αλλά η Κομισιόν πρέπει να μας δείξει πού είναι καλύτερο να δοθούν τα χρήματα ώστε να εξυπηρετούν περισσότερο και καλύτερα τους στόχους μας και να μην καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερος που η Επιτροπή Προπολογισμών παίζει σημαντικό ρόλο και στον καθορισμό αυτής της πολιτικής. Τώρα. Ευχαριστώ, συγκητή. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα, μετά την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων, η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 29 Μαΐου της Αλώσεως και στην Επιτροπή μας θα εγκριθεί η γνωμοδότηση 20 Ιουνίου διότι η Επιτροπή Αλληλείας προβλέπει την έγκριση της έκθεσής της στις 10 και 11 Ιουλίου για ψηφοφορία στην Ολομέλεια μετά. Να αυτά. Το σημείο 7. Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα. Ο κύριος Έπινγκ είναι ο συντάκτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος που θα δώσει το πλαίσιο για να αναπτυχθεί, να παραχθεί και να διαδοθεί το σύνολο των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για την περίοδο 2013-2017. Το συνολικό ποσό είναι 299,4 εκατομμύρια ευρώ για την πενταετία του προγράμματος συμπεριλαμβανομένων και των 57,3 εκατομμυρίων για την προηγούμενη περίοδο, ενώ τα υπόλοιπα από τα 299 είναι για την περίοδο 2014-2017. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, ESS, είναι συνεργασία της Eurostat με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες ή Αρχές και αντιμετώπισε προκλήσεις και δυσκολίες το τελευταίο διάστημα περιλαμβανομένης και της ανάγκης ευρωπαϊκών στατιστικών και της αλλαγής του τρόπου με τον οποίο συλλέγονται τα στοιχεία όταν έχουμε και περικοπές στους εθνικούς και στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ποιος είναι ο βασικός στόχος. Να μπορεί το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα να είναι ο βασικός πάροχος υψηλής ποιότητας στατιστικών στην Ευρώπη. Τρεις είναι οι γενικοί στόχοι κανονικά σε όλες τις δράσεις. Ποιοτικά στατιστικά στοιχεία, το πρώτο. Το δεύτερο, νέες μέθοδοι ε, για να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποδοτικότητα και το τρίτο να ενισχυθεί η σχέση της ε, Ευρωπαϊκής ε, Στατιστικής Αρχής με τις εθνικές για να αυξηθεί η παρεγωγικότητα. Για να γίνουν όλα αυτά θα εγκρίνεται κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέτει τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι τροπολογίες μου αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή χρηματοοικονομική κρίση επιδεινώθηκε πολύ γιατί δεν είχαμε έγκαιρα, ε, ε, ακριβή και υψηλής ποιότητα στατιστικά στοιχεία. Γι' αυτό έχω κάνει τροπολογίες που τονίζουν την ανάγκη ε, να έχουμε διαρκώς ε, ακριβή στοιχεία που να προέρχονται από ανεξάρτητες εθνικές στατιστικές αρχές με τους αντίστοιχους και σωστούς μηχανισμούς ελέγχου και ε, εποπτείας για να μην έχουμε υπολειτουργία και υποπαραγωγικότητα για λόγους ρουτίνας. Τα ακριβή στατιστικά στοιχεία είναι απολύτως ουσιώδη για να διατηρηθεί το σημερινό ευρωσύστημα θα ήθελα να σας παραπέμψω στις πολιτικές του Sir John Κόπερτρέιτ, πρώην ε, ε, υπεύθυνο ε, για τα οικονομικά στο Hong Kong από το 61 μέχρι το 71 που ήταν η θετική μη παρέμβαση το πρόγραμμά του και το Hong Kong έγινε ένα πολύ εύρωστο οικονομικό κέντρο παγκοσμίως. Αυξήθηκε κατά 50% το εισόδημα, η μισθή και μειώθηκε κατά 2 τρίτα η φτώχεια. εμεί, ούτε να το ενερευόμαστε δεν μπορούμε αυτό. Και ο Σερ Τζον ε, βάσισε το πρόγραμμά του στι σωστέ οικονομικέ στατιστικέ. Και όταν το ρώτησαν τι θα πρέπει να κάνουν φτωχέ χώρε, ένα πράγμα απάντησε να καταργήσουν την εθνική του στατιστική υπηρεσία. Αυτή ήταν η συμβουλή που έδινε ο Σερ Τζον σε εκείνου που σχεδίαζαν τι οικονομικέ πολιτικέ. Ωραία αυτά τα ιστορικά στιγμιότυπα. Δεν ξέρω εάν ε, συμφωνούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Καλύτερα να είμαστε προμηθείς παρά επιμηθείς νομίζω και να φροντίζουμε εκ των προτέρων να διορθώσουμε τα πράγματα είτε το κάνουμε αυτό για τους σωστούς είτε για τους λάθος λόγους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σεγητά. Συγχαρητήρια. Σε συγχαίρω λοιπόν γιατί μας κάνατε να χαμογελάσουμε γύρω από θέματα σοβαρά δηλαδή στατιστικά. Ήταν αξιόλογο αυτό το οποίο είπατε. Στην ίσο του Χονγκ Κόγκ οι στατιστικές ε, δεν υπήρχαν τη δεκαετία του 70 με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Γιούτε θέλει το λόγο για την πολιτική ζωή στο Χονγκ Κόγκ, μήπως όχι. Ο κύριος Γκάιερ όμως έχει ζητήσει το λόγο για την πολιτική ζωή και την οικονομική στο Χονγκ Κόνγκ δυστυχώς δεν έχω άποψη, αλλά στη Γερμανία είναι πολύ γνωστό ε, αυτό που είχε πει ο Winston Churchill κάποτε. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ καμιά στατιστική που δεν την έχεις να θεύσει εσύ ο ίδιος. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Έχουμε όλοι η προσωπική εμπειρία και εδώ στην Επιτροπή μας. Γνωρίσαμε τα προβλήματα ακριβώς ε, λόγω της ε, μη σωστής ε, συλλογής στατιστικών στοιχείων. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας για να μπορεί να ασκεί μια λογική πολιτική και ένα σχεδιασμό με βάση αξιόπιστα στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής. Γι' αυτό Θεωρώ πολύ σημαντικό να συνεργάζονται οι υπηρεσίες μεταξύ τους και ε, οι στατιστικές αρχές. Και επίσης σημαντικότερο να είναι ανεξάρτητες. Γιατί έχουμε πάλι κακιά πείρα από το παρελθόν με την έλλειψη ανεξαρτησίας τέτοιων ε, υπηρεσιών. Ακριβώς επειδή ισχύουν αυτά όμως, έχω προβλήματα εγώ. Για να συμφωνήσω με την έκθεση του κυρίου Έπινγκ. Πώς να το πω. Με την ιδέα ότι θέλει να κάνει και οικονομία. Εμείς κάνουμε αυτή τη συζήτηση για όλα τα προγράμματα που μπορούμε να έχουμε περικοπές στους προπολογισμού. Αλλά ε, αυτό είναι και το πολιτικό πιστεύω της πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκει ο κύριος Έπινγκ. Όταν λέμε όμως ότι είναι τόσο σημαντικό όλα αυτά, να έχουμε καλά στατιστικά στοιχεία για να κάνουμε σωστή ε, πολιτική και προγραμματισμό και σχεδιασμό, ε, δεν μπορούμε μετά να ερχόμαστε και να λέμε αν μειωθεί και ο προπολογισμό. Είναι σαν τις 10 εντολές. Ότι θα πρέπει πάντα, λέμε, να είμαστε φρόνιμοι και συνεπείς και φιδωλοί. Είμαι ο τελευταίος που θα το κρούσω αυτό ως ε, μέλος Επιτροπής Προϋπολογισμών. Αλλά ε, το να κάνουμε εδώ οικονομίες είναι πραγματικά σε λάθος τόπο οικονομία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάτσνη έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είμαι σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ. Και πράγματι στις στατιστικές πολλές φορές ε, περιλαμβάνονται σοφά πράγματα και ελπίζω να μην ε, μετατρέπονται συχνά σε ψεύδι αυτά τα θαύματα. Πάντως καλό είναι να υπογραμμίσουμε μέσω των στατιστικών ότι μέσω των στατιστικών πετυχαίνουμε τη σωστή αξιολόγηση των πολιτικών μας. Είναι απαραίτητο λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία και γι' αυτό θα συμφωνήσω με τον εισηγητή και με τους στόχους τους οποίους θέτει έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν οι στατιστικές τα υπάρχοντα στοιχεία, τα ισχύουσες καταστάσεις και είναι σωστή η έκκληση για βελτιώσεις και για αύξηση της παραγωγικότητας μέσω εταιρικών συνεργασιών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ από πλευράς της πολιτικής μου ομάδας θα παρακολουθήσω το θέμα αυτό και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία να είναι αποδεκτή από τη μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και η οποία να μπορέσει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμεθα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Στάτσνη. Κοιτάξτε, έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται τεχνικής φύσεως, αλλά έχει όμως ε, θέτει διακυβεύματα οικονομικά και πολιτικά σημαντικά. Σε μια χώρα σαν τη δική μου, που δεν είναι από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο βέβαια, δεν αναγνωρίζουμε το επίπεδο βιομηχανικής και οικονομικής παραγωγής παρά μόνο με καθυστέρηση τριών μηνών, γιατί το σύστημα συλλογής των στοιχείων βασίζεται σε επαγγελματικές οργανώσεις, ανακλάδο βιομηχανικό και είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό και αργό. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε προβλέψεις σχετικά αξιόπιστες για το επίπεδο της ανάκαμψης σε έξι μήνες ή σε ένα χρόνο, εάν δεν γνωρίζουμε, εάν πριν τρεις μήνες η βιομηχανία βρισκόταν σε ύφεση ή σε ανάκαμψη. Τουλάχιστον με τη λεγόμενη μετεωρολογία μπορούμε να πούμε αν σήμερα βρέχει. Με τη στατιστική όμως δεν μπορούμε να πούμε παρά θα ξέρουμε σε τρεις μήνες αν στη γαλλική βιομηχανία τα πράγματα πηγαίνουν καλά ή όχι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα στατιστικά μας μέσα είναι ουσιαστικά χρήσιμα για την σωστή διακυβέρνηση της οικονομικής πολιτικής και τη στιγμή κατά την οποία υπό την πίεση της κρίσης τα κράτη-μέλη μας ενισχύουν την δημοσιονομική συνεργασία και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και για 25 χώρες από τις 27 στη Νέα Συνθήκη, έτσι ώστε οι οικονομικές πολιτικές να εναρμονιστούν καλύτερα μεταξύ τους, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ε, το θετικό του τμήματος και να μεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη, είναι απαραίτητα τα στατιστικά στοιχεία. Ξεκινήσαμε σήμερα μιλώντας για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και για τα αναγκαία επίπεδα και διαπιστώνουμε ότι επί τη βάση ε, θα έλεγα των στοιχείων στα οποία στηρίζουμε την πολιτική μας τα τεχνικά μας μέσα εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή και χρήζουν βελτίωσης. Αυτά όλα λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε πιο προσεκτικά. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Έπινγκ Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία για τις τροπολογίες στην έκθεση ΕΠΕΝ είναι η 14η Μαΐου, επόμενος μήνας δηλαδή. Θα πρέπει να θέσουμε σε ψηφοφορία τη γνωμοθότησή του στις 31 Μαΐου και σε επίπεδο θα έλεγα βασικής πρόβλεψης και πρέπει να επιβεβαιωθεί στις 18 Ιουνίου η Επιτροπή ΕΚΟΝ που είναι η αρμόδια επί της ουσίας θα ψηφίσει την έκθεσή του. Αυτά μπορούμε να περάσουμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Φάσμον για τη δημιουργία ενός προγράμματος δράσης για τα τελωνία και τα φορολογικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυτό το σύστημα για να αντικαταστήσει το πρόγραμμα Customs Τελωνία 2013 και Fiscalis 2013. Αυτό ονομάζεται τώρα Fiscus και συμμετέχει και στο με στόχο να ε, απλουστευτεί όλη αυτή η προσπάθεια υποστηρίζει τα τελωνία ε, και είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Customs 2013, ενώ σε αντίθεση το 2013 Fiscalis ε, στόχο έχει να ενισχύσει την ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να συνεργάζονται καλύτερα οι φορολογικές υπηρεσίες και τα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία των κρατών μελών. Είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα το οποίο δεν μπαίνει στα χωράφια όμως της φορολογικής πολιτικής που κατά κύριο λόγο είναι η αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, δεν μπορούν τα δύο προγράμματα όμως να ε, συγχωνευτούν ως προς τη νομική τους βάση. Έχω επιφυλάξει σε αυτό. υπάρχει πρόβλημα για την εφαρμογή, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση. Επιπλέον, ε, καμία από τις δύο ε, προτάσεις για ενδιάμεση αναθεώρηση δεν προσφέρονται και παρά τη αιτιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι σωστό να συγχωνευθούν τα δύο προγράμματα, τα οποία λειτουργούν πολύ καλά ως ξεχωριστά αυτοτελή προγράμματα, σύμφωνα με τις ε, αξιολογήσεις που έχουν κάνει οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι. Επιπλέον, από τότε, ε, μάλλον εφόσον έχει διαφορετική πρικοδότηση προβλέψει για τα δύο προγράμματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλει να διατηρηθεί και ταυτότητα των προγραμμάτων, θα φαινόταν λογικό ότι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί αυτό θα ήταν να παραμένουν χωριστά τα προγράμματα. Υποστηρίζω πλήρως ε, και τα δύο προγράμματα, και το Fiscalis και το Customs, αλλά θα πρότεινα ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σκεφτεί είτε να απορρίψει την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε οι καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου να προτείνουν άλλη δράση και τελικά δύο ξεχωριστές νομικές βάσεις για κάθε πρόγραμμα. Μία. Αυτό θα επιτρέψει ε, να ε, συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά με το σωστό τρόπο τα δύο προγράμματα. Αυτή τη θέση την ακολουθούν και οι Επιτροπές Οικονομικών και Νομισματικών ε, Υποθέσεων και Εσωτερικής Αγοράς και στις 18 Απριλίου επίσης η ε, διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών μετά από αίτημα των Επιτροπών ΕΚΟΝ και ΙΜΚΟ. Δίδεται λοιπόν ε, μια νέα ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει τι θέλει Μάλλον έγινε αυτό στη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών, αλλά ε, δεν ε, μας έπεισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα θα δούμε κατά πόσο θα κληθούμε να εφαρμοστούμε το άρθρο 51 του κανονισμού. Προς ενημέρωσή σας, η Γραμματεία ενημερώθηκε από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου ότι υπήρχαν και κάποιες επιφυλάξεις ε, για το κατά πόσο στο νομοθετικό κείμενο είναι παραδεκτές ορισμένες από τις δικές μου προτάσεις. Έχω κάνει όμως συζητήσεις με την γραμματεία και οι τροπολογίες 1, 3 και 4 στοχεύουν να δώσουν ένα πολιτικό μήνυμα στις καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές και δεν φιλοδοξούν ε, στο να εγκριθούν ως νομοθετικό κείμενο από την Ολομέλεια. Προσβλέπω συνεργασία με τους σκιώδεις ηγητές για τη γνωμοδότηση και παραμένω στη διάθεσή σας ε, για περαιτέρω τροπολογίες εξ των πολιτικών ομάδων και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε ο κύριο Στόλογιαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ το συντάκτη γνωμοδότησης. Ε, όντως, είναι δύο οι καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές, επί της ουσίας δηλαδή ΕΚΟΝ και ΙΜΚΟ, βάσει του άρθρο 51 του κανονισμού, και οι δύο πρόεδροι των δύο επιτροπών απίφθηναν επιστολή στο Συμβούλιο για να υπογραμμιστεί η ανάγκη να διαχωριστεί το πρόγραμμα φίσκους σε δύο προγράμματα, όπως ίσχυε στο παρελθόν. Ένα για τα τελωνία και ένα άλλο για τα φορολογικά ζητήματα. Στις 16 Μαΐου η διάσκεψη των Προέδρων συνεδριάζει και αναμένουμε να εγκρίνει αυτή την αποστολή που έχουν υπογράψει οι Πρόεδροι των δύο Επιτροπών, Οικονομικών Υποθέσεων και Εσωτερικής Αγοράς. Η αποστολή, μάλλον η επιστολή αυτή θα αποστολή στο Συμβούλιο και την αναμένει το Συμβούλιο για να κανονίσει την πορεία του από εκεί και πέρα. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του εισηγητού, βεβαίως και συμφωνούμε με την τροπολογία να σπάσει αυτό το πρόγραμμα στα δύο και επίσης υπάρχει και μια άλλη τροπολογία που τονίζει ότι η χρηματοδότηση που ορίζεται από αυτή την νομοθετική πρόταση είναι ενδεικτική και μόνο προς την νομοθετική αρχή και δεν μπορεί να οριστεί μέχρι να συμφωνηθεί η πρόταση για ένα κανονισμό που θα ορίζει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2020. Και εμείς υποστηρίζουμε και αυτή την τροπολογία γιατί θεωρούμε λογική. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο, όπως είπε ο εισηγητής μας προηγουμένως. Α, όχι, ο κύριος Γκάιερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι σκιώδης ηγητής για τους σοσιαλδημοκράτες. Και θα ήθελα παρακαλώ εδώ να ρωτήσω κάτι στις πολιτικές ομάδες. Είναι πραγματικά απαραίτητο να χωριστούν τα δύο προγράμματα. Έχω καταλάβει ότι η φορολογία και το τελωνίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες έχουν διαφορετικό καθεστώς. Εντάξει, αυτό όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να υπερισχύσει ως επιχείρημα. Γιατί αυτό άκουσα. Ε, για να χωριστεί και πάλι το πρόγραμμα. Δεν έχω καταλάβει γιατί ισχύει αυτό το επιχείρημα. Γιατί και στους δύο τομείς πρόκειται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Δηλαδή και στα δύο έχουμε έσοδα για τον προϋπολογισμό που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα και αν ε, τα έσοδα από τα τελωνία και τα έσοδα από τη φορολογία συνενωθούν, τότε μπορούμε να μειώσουμε και τις εθνικές συνεισφορές στον κοινοτικό προϋπολογισμό για να κάνουμε και ένα βήμα προς την κατεύθυνση των κυβερνήσεων που ζητούν να μειωθεί η συνεισφορά τους. Δεν είναι δική μου θέση, δεν την υιοθετώ αυτή απόλυτα, αλλά είναι και αυτό ένα επιχείρημα. Και θα με εξέπλητε αν το κοινοβούλιο εδώ εκπροσωπούσε μια θέση που λέγει ότι δεν συμφωνούμε με το, αυτό το πιο αποτελεσματικό μέσο για λόγους τυπικούς. Να το χωρίσουμε σε δύο προγράμματα και να διακυβευτεί η δυνατότητα συλλογής περισσότερων εσόδων. Γιατί εγώ ξέρω μερικά που ε, οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την ποινική δίωξη για αδικήματα στα τελωνία είναι οι ίδιες που αφορούν και τις φορολογικές ε, ποινικέ υποθέσεις. Και έτσι τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση καλύτερα να ανταποκρίνονται και στο καθήκον τους και να διαφυλάτουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό και συνεπές. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής θέλει ξανά το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Εμείς δεν θέλουμε να διαιρέσουμε το πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε με το παρόν πλαίσιο, να συνεχιστεί δηλαδή το α, καθεστώς το οποίο ισχύει σήμερα. και η αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας άλλωστε συστήνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό που σας ζήτησα και εγώ. Και νομίζω ότι πίσω από την πρόταση αυτή υπάρχει μια κάποια συνένεση. Bon. Très bien. Donc, je suppose qu'il y aura d'autres amendements. Σε ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα υποθέσω ότι υπάρχουν και άλλες τροπολογίες. Όπως το είπε ο εισηγητής μας, κάποιες από τις δικές του τροπολογίες προκάλεσαν κάποιες επιφυλάξεις από πλευράς των υπηρεσιών κατάθεσης τροπολογιών για το αποδεκτό ή μη. Πρόκειται για τις τροπολογίες οι οποίες συνδέονται με την ύπαρξη των προβλημάτων στα οποία αναφερθήκαμε για την ύπαρξη ενός προγράμματος ή δύο προγραμμάτων. Πράγματι, σε επίπεδο ολομέλειας θα τεθεί το θέμα επί τη βάση του κειμένου των τροπολογιών που θα έχουν ε, δεχτεί ήδη οι επί ε, ε, επιτροπές και όχι η Επιτροπή μας. Ναι. Η Επιτροπή μας μπορεί να καταθέσει τροπολογίες ακόμα και αν δεν τις θεωρεί αποδεκτές η υπηρεσία της Ολομέλειας. Αντίθετα με τις Επιτροπές επί οι οποίες θα πρέπει να αποφασίσουν ποιες ε, ε, τροπολογίες θα κατατεθούν στην Ολομέλεια ή μη. Όπως είπε ο εισηγητής υπάρχουν δύο διαφορετικές επί της ουσίας επιτροπές, η ΙΝΚΟ και η ΕΚΟΝ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι 23η Μαΐου με στόχο την ε, υιοθέτηση της νομοδότησης την 21η Ιουνίου. Καλώς λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Με το σημείο 10. 9 πρώτα, όχι λάθος λέω ο πρόεδρος, το σημείο 9. Πρόκειται για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής του Ταμείου λοιπόν Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Ο κύριος Ιάν Κοσλόφσκι έχει ζητήσει το λόγο, είναι ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στοχεύει να βοηθάει στους εργαζόμενους που δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές. 500 εκατομμύρια είναι το ανώτα, είναι ο προϋπολογισμός του και προβλέπεται ότι δεν μπορεί να ξεπερνάει το 0,35% του γενικού προϋπολογισμού, δηλαδή 1.700.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή Υπάρχει το σύνολο του ποσού αυτού. Η Κομισιόν στις 4 Απριλίου υπέβαλε την πρόταση απελευθέρωσης του 1.120.000 για την τεχνική βοήθεια. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μείνουν 630.000 στο αποθεματικό για επίγουσα περίπτωση παρέμβασης. Τα ποσά αυτά θα κατανεμηθούν λέει ως εξής. Εποπτεία, συντήρηση στο σελίδων, εκτύπωση υλικού και ετησίων εκθέσεων, και πληροφόρηση για την καλύτερη δυνατή χρήση, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, δικτύωση και προετοιμασία της τελικής αξιολόγησης από εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Το αίτημα της Κομισιόν συμφωνεί με τα ισχύοντα, με τον κανονισμό δηλαδή λειτουργίας του Ταμείου αυτού. Γι' αυτό βρίσκω περίεργο ότι μερικές χώρες μέλη αντιτάχθηκαν στην απελευθέρωση του διάθεση του ποσού αυτού. Το Συμβούλιο αποφάσισε να παγώσει την εξαίρεση για την αντιμετώπιση της κρίσης για να βοη... που στόχευε στη βοήθεια των εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους ή που γενικά βλάφτηκαν από την παγκοσμιαποίηση ενώ αυτό ήταν μέχρι από την αρχή ένα βασικό στοιχείο αλληλεγγύης και γι' αυτό ζητώ από το Συμβούλιο <coughs> να αλλάξει γνώμη. Για να συνοψίσω, στον φετινό προϋπολογισμό οι πληρωμές για το ταμείο αυτό χορηγήθηκαν από χωριστή γραμμή του προπολογισμού. Αυτό ζητούσαμε ανέκαθεν ως κοινοβούλιο γιατί το ταμείο αυτό είναι ανεξάρτητο εργαλείο και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με άλλες θέσεις, με δική του θέση να προβλέπονται τα πόσα. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά, κύριε Βέρντεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ μιλώ ως σκιώδης της ομάδας μου των σοσιαλιστών και ως μέλος της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Απασχόλησης. Τρία σημεία. Πρώτον, όπως μάλλον ξέρετε, η ομάδα εργασίας αποφάσισε να τροποποιήσει λιγουλάκι την μέθοδο εργασίας της, δηλαδή να υποβάλει τροπολογίας οι οποίες θα αναφέρουν το περιεχόμενο της επιστολής σύμφωνα με αυτά που είπε και ο εισηγητής. Τι τροπολογίες είναι αυτές λοιπόν. Καταρχήν εκφράζουμε τη λύπη μας για γιατί δεν έγινε η τελική αξιολόγηση που χρηματοδοτείται ακριβώς από αυτή την τεχνική βοήθεια. Αναρωτιόμαστε για τις επιπτώσεις θετικές ή όχι που είχε αυτή η τεχνική βοήθεια. Υπενθυμίζουμε την ανάγκη να επιταχυνθεί η κινητοποίηση και τέλος στηρίζουμε τη χρηματοδότηση μιας ομάδας επαφών ή εμπειρογνωμόνων μέσω της χορήγησης κονδυλίων τεχνικής βοηθείας ακριβώς. Συμφωνώ γενικά με τον εισηγητή, ιδίως ως προς τη σημασία που έχει το ταμείο αυτό και τελευταίο η έγκριση αυτού του ποσού για την τεχνική βοήθεια δεν έγινε από το Συμβούλιο λόγω μιας μειοψηφίας που το θεώρησε το ποσό αυτό υπερβολικά υψηλό σε σύγκριση με το 11 αλλά το επιχείρημα αυτό δεν μου φαίνεται σωστό κατ' εμέ είναι πρόφαση για να δυσκολευτούν ακόμη περισσότερα τα πράγματα για το ταμείο αυτό. Ευχαριστούμε κύριος Χάγκελουντ. Στη δική μας ομάδα, Πρόεδρε, θέλουμε να υπάρχουν επαρκή κονδύλια για το ταμείο αυτό. Είτε πρόκειται για τους στόχους που είχαμε θέσει, είτε για να συμφωνούμε με αυτά που είχαμε πει από την αρχή. new Τώρα βέβαια δεν συμφωνούν όλοι με το κόστος που αντιπροσωπεύει η κινητοποίηση του ποσού και γι' αυτό παρά το ότι είναι, υπάρχουν και θετικά στοιχεία στην πρόταση εμείς δεν τη δεχόμαστε τελικά. Ευχαριστούμε πολύ. Από αυτά που είπε ο κύριος Ντάρντεν λοιπόν συμπεραίνω ότι η Επιτροπή Απασχόλησης δεν θα μας στείλει μόνο χρωμοδότηση αλλά και ντροπολογίες. Λόγω δε των διοριών που έχουμε, προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος, στις 30 Μαΐου θα εγκριθεί η γνωμοδότηση εκείνη και εμείς θα τοποθετηθούμε την επομένη στις 31. Πρέπει λοιπόν η τροπολογία, αυτή η τροπολογία είναι γραμμένη σε μία από τις μεγάλες γλώσσες της Ένωσης και μάλιστα σε εκείνη με την οποία εργαζόμαστε συνηθέστερα. Ένας Γάλλος λέει στα φλαμανδικά ή στα βαλονικά. Όχι, όχι, αυτό είναι δύσκολο. Όχι, δύσκολο. Όχι, νομίζω θα μπορέσει να μεταφραστεί γρήγορα σε όλες τις γλώσσες μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο εισηγητή. Το θέμα αυτό σχετίζεται και με τη μεταφορά που θα ψηφίσουμε σε λίγο, την υπαριθμόν 3 δηλαδή. Η προθεσμία διαδόση των προγειών στην Επιτροπή μας λήγει στις 16 Μαΐου το μεσημέρι. 30 Μαΐου θα, θα ψηφίσει άλλη Επιτροπή και εμείς τέλη Μαΐου και μετά στην Ολομέλεια 12 και 13 Ιουνίου. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας κύριο Κοζηλόφσκι. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή του σημείου 10. Το πρόγραμμα Καταναλωτές για την περίοδο 14-20 των Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εκατομμύρια καταναλωτών και ότι πρόκειται για ένα 56% του ΑΕΠ και το, πρόγραμμα για το 2014-2020 είναι περιορισμένο. 197 ε, εκατομμύρια ευρώ και 20,7 είναι για διοικητικές δαπάνες. Στόχος είναι να μπει ο καταναλωτής στο επίκεντρο ε, της ενίας αγοράς και να μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του και να τα απολαμβάνει αυτό δεν θα πρέπει να είναι αυτόνομος ξεχωριστός στόχος, αλλά ένα στόχος ενιαίος γενικά που να διαπερνά όλες τις πολιτικές, τους τέσσερις στόχους που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασφάλεια, πληροφόρηση και εκπαίδευση, δικαιώματα και ένομη προστασία και επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας. Αυτές είναι οι τέσσερις προτεραιότητες, οι τέσσερις στόχοι. Βεβαίως είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση και δυνατότητα αυτών των δικαιωμάτων, καθώς επίσης είναι πολύ σημαντική και η δυνατότητα προσφυγής ε, που πρέπει να έχουν οι καταναλωτές. Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη τους θα ήταν θετικό να δημιουργήσουμε ένα κέντρο, ένα ευρωπαϊκό κέντρο πιστοποίηση για τις επιγραμμικές πωλήσει και τις εταιρείε που πολλούν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο και να υπάρχουν σωστοί στατιστικοί δείκτες. Είναι γελίο να χρησιμοποιείται ως δείκτης για την εύρυθμη λειτουργία μιας αγοράς ο αριθμός των παραπώνων και καταγγελιών. Δηλαδή αν δεν έχουμε καμία καταγγελία είναι 100% σωστή αγορά και λειτουργεί εύρυθμα. Μα δεν μπορεί να είναι αυτός ο δείκτης για την αξιολόγηση. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός δείκτης και ο μοναδικός τρόπος ε, επαλήθευση αν λειτουργεί σωστά μια αγορά. Οπότε, θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση, να υπάρχει ε, και συμφωνία και συνένεση ως προς τους δείκτες. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τις καταγγελίες και να ε, τις προσπηγές τους ε, ως ε, φυσικά πρόσωπα χωρίς να ανήκουν σε μια ένωση προστασίας των καταναλωτών. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις ενώσεις, δεν αντιλέγω, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ένας μεμονωμένος καταναλωτής να μπορεί κάπου να προσφεύγει, να χρησιμοποιεί όλα τα ηλεκτρονικά ένωμα μέσα με τρόπο εύκολο, χωρίς να είναι μέλος μιας ένωσης καταναλωτών. Και όχι μόνο εύκολο, αλλά και όχι δαπανηρό. Γι' αυτό προτείνω να υπάρχει ένας οργανισμός, ένα κέντρο, πάση περιπτώσει, ενιαίο και να μπορούν να προσφεύγουν όλοι οι καταναλωτές και να μοιράζονται τα παράποντα και τις καταγγελίες τους. Μια πλατφόρμα έτσι διαδραστική. για να προωθούνται και βέλτιστες πρακτικές. Όλα αυτά ε, τα γράφω και στις τροπολογίες μου. Αλλά νομίζω ότι γενικά συμφωνούμε. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Φέρμα. Μια σύντομη σκέψη. Ο σκιώδης εισηγητής της ομάδας μου δεν είναι παρόν. Για τις τροπολογίες 2 και 3. Στην τροπολογία 2 ο εισηγητής αναφέρει, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα σε ποσά, αλλά λέει ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι χαμηλή. Και εδώ αφήνει να εννοηθεί ότι προτιμά μια διαφορετική ανώτερη τιμή. Στην τροπολογία 3 λέει επίσης ότι οι δικαιτικές δαπάνες είναι πολύ υψηλές και ζητά την Επιτροπή να δικαιολογήσει και να επανεξετάσει τις δαπάνες αυτές. Δεν ξέρω, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα γενικό πρόβλημα. Όλο και περισσότερες δαπάνες ζητάμε εμείς και περιμένουμε διοικητικά να μειωθούν τα κόστη. Αυτή η λογική δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα καθυστερήσεων, εφαρμοστικά προβλήματα και προβλήματα απλά εκτέλεσης κάποιων διοικητικών δαπανών που είναι απαραίτητες να υπάρξουν γιατί αλλιώς δεν θα λειτουργήσουν τα προγράμματα. Και γι' αυτό θα ήθελα ο εισηγητής να εξετάσει προσεκτικά τη συγκεκριμένη περίπτωση, να σας πει αν πράγματι για το πρόγραμμα αυτό υπάρχει πράγματι μια γενναιόδορη διοικητική ε, πίστοση, αλλιώς να είμαστε πιο προσεκτικοί. Η Αντιπρόεδρος, η κυρία Χάουγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κατανοώ αυτό. Αλλά ακριβώς αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μικρά τα προγράμματα. Όχι μόνο αυτό για την προστασία των καταναλωτών, θα το βρούμε μπροστά μας και αλλού. Στο πρόγραμμα δράσης για την υγεία. Είναι λίγα-λίγα μικρά προγράμματα που θα πρέπει να τα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ είμαι η τελευταία που θα υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διοικητικές δαπάνες. Αλλά εδώ πραγματικά, αν δεν τους δώσουμε τα κονδύλια, δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα. Και τελικά θα έρθουμε να αναρωτηθούμε και θα ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν θα εφαρμόστε. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτό το μικρό πρόγραμμα που δεν υπάρχει καν σε διαχείριση. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη αρμόδια διοίκηση, υπηρεσία να το κάνει. Όλα πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και καλά το κάνει και το θέλουμε, αλλά θα πρέπει να τις δώσουμε και τα μέσα. Merci, ε, Monsieur... Ευχαριστώ, Ιούτα. Θέλει να απαντήσει ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει εδώ καμία ε, αναντιστοιχία όταν λέω ότι είναι μικρό το πρόγραμμα ή χαμηλή η πρικοδότηση, δεν σημαίνει ότι ζητώ ταυτόχρονα περισσότερα κονδύλια. Αλλά σκεφτούμε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη είναι 500 εκατομμύρια και από πλευρά ΑΕΠ αυτό αντιπροσωπεύει ένα 56%. Αν δεν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι με ένα πρόγραμμα που θα έχει πραγματική θέση στην αγορά και θα ενημερώνει τους καταναλωτές, είμαι πεπισμένος ότι αυτό το ποσό δεν επαρκεί. Για τους στόχους. Σας λέω ότι είναι χαμηλό το ποσό. Αν θέλετε εγώ να αναθεωρήσω τον όρο που χρησιμοποιώ. Είπα ότι είναι χαμηλό το ποσό γιατί θεωρώ ότι είναι χαμηλό και θα πρέπει να μας προβληματίσει. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι χαμηλό τι να σας πω. Οι διοικητικέ δαπάνες είναι πάνω από 10% στο πρόγραμμα. Αλλά στις διοικητικέ δαπάνες δεν ζητώ περικοπές. Αυτό που λέγω είναι ότι θα πρέπει να τις δικαιολογήσουν και να τις αναθεωρήσουν, επανεκτιμήσουν. Αλλά με περικοπή δεν συμφωνώ. Γιατί αυτό θα υπονομεύσει το ίδιο το πρόγραμμα, την εκτέλεσή του ή του στόχους του. Που σας είπα είναι 197 εκατομμύρια. Που είναι χαμηλό ποσό. Είναι λίγα τα χρήματα και το 20, τα 20,75 εκατομμύρια είναι διοικητικές δαπάνες. Γι' αυτό σε μία από τις τροπολογίες μου λέγω ότι θα πρέπει ενδεχομένως να προχωρήσουμε προς ε, ένα εκτελεστικό ε, φορέα, οργανισμό, έτσι ώστε να υπάρχουν πλέον εκτήματα και να γίνει μια εξάρτητη ανάλυση κόστους-οφέλους που θα αποδείξει ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα. Όντως, γύρω από το συγκεκριμένο πρόγραμμα τώρα, η ανταλλαγή απόψεων έδειξε ένα πρόβλημα γενικότερο την σχέση ανάμεσα σε λειτουργικές δαπάνες και διοικητικές δαπάνες. Αυτό θα τεθεί περισσότερο ακόμα και σε άλλα προγράμματα και αυτό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα της δημοσιονομικής διαπραγμάτευσης του επόμενου πολυετούς προγραμματισμού, όχι μόνο στην κατηγορία 5, αλλά κάτω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τις λειτουργικές πιστώσεις. Αυτό τίθεται και σε επίπεδο εξωτερικών υπηρεσιών, ισχύει και για τις υπόλοιπες πολιτικές, υπάρχει ο κίνδυνος πολύ υψηλών διοικητικών δαπανών, υπάρχει όμως και ο κίνδυνος του να μην υπάρχουν αρκετές δαπάνες. Mm. Ένας Άγγλος κοινωνιολόγος, ο Ρότς Πάρκινσον, ο οποίος είχε πει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μελετώντας τις εξελίξεις στο προσωπικό και στα πληρώματα του βασιλικού ναυτικού σε εποχές ειρήνης και είχε πει ότι το προσωπικό ε, σε εποχές ειρήνης ήταν περισσότερο από ό,τι σε εποχές πολέμου. Και όσο λιγότερα πλοία υπήρχαν και όσο λιγότεροι ναύτες υπήρχαν, τόσο περισσότεροι υπάλληλοι υπήρχαν διοικητικοί στα Υπουργεία γιατί ασχολιόντουσαν με τους αναπήρους, τους εφέδρους, τους υπαλλήλους κτλ. Στη Γαλλία, πιο κοντά σε εμά, οι αστυνομικές υπηρεσίες πρόσφατα είχαν περισσότερους υπαλλήλους στις δικητικές τους υπηρεσίες παρά στους δρόμους για να διασφαλίσουν την αστυνόμευση και την ασφάλεια των πολιτών. Όταν λοιπόν κάνει κανείς τέτοιες συγκρίσεις ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών βλέπει ότι η σχέση ανάμεσα στους διοικητικούς υπαλλήλους με τους εκπαιδευτικούς ποικίλει από ένα με δύο σε, ε, σε διάφορες χώρες. Λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος για υψηλές διοικητικές δαπάνες. Υπάρχει όμως και ο αντίθετος κίνδυνος, η μείωση των διοικητικών δαπανών σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να μην είμαστε σε θέση πλέον να ασκήσουμε τις πολιτικές και να χρησιμοποιήσουμε τις λειτουργικές πιστώσεις με ικανοποιητικό τρόπο. Είναι λοιπόν το θέμα αυτό σημαντικό και πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά όπως το κάνει ο εισηγητής μας για το πρόγραμμα καταναλωτής. Για το χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 14η ε, Μαΐου μεσημέρι. Η συζήτηση θα γίνει στις 31 Μαΐου και η ψηφοφορία στην ΙΝΚΟ επί της ουσίας θα γίνει την 20η Ιουνίου έτσι ώστε να φτάσει στην Ολομέλεια της 12ης Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ τον εισηγητή και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Νιένσκι για τα 11 και 12 και εδώ πρέπει να εκφέρουμε γνωμοδοτήσεις ε, για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Κυρία Νιένσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να αναφερθώ στη γνωμοδότηση που συζητήσαμε. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό για τη βοήθειά του στην προετοιμασία αυτής της γνωμοδότησης. Αυτοί οι κανόνες για τις διαδικασίες εφαρμογή μηχανισμών κεντρικής ένωσης της δράσης είναι ένα πλαίσιο που αποτελεί κάτι το τελείως καινούργιο και που ελπίζουμε να μας δώσει μεγαλύτερη διαφάνεια για τις δαπάνες για εξωτερικές δράσεις επίσης, ενώ και η παραμικρότερη δεκάρα πρέπει να συμφωνεί με το πρόγραμμα πλαίσιο προβλέπονται και εξαιρέσεις από τους κανόνες. Και γιατί αυτό, γιατί αυτό. Πολύ απλά, γιατί οι εξωτερικές δράσεις διαφέρουν πολύ από τις εσωτερικές, διότι έχουν διαφορετικούς στόχους για να στηρίξουν πολύ διαφορετικά ρικές συνθήκες σε σύγκριση με το κανονική λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου. Πρέπει λοιπόν να επιτηρούμε τη σωστή του χρήση και το εργαλείο καλής γειτονίας, εξωτερικής βοηθείας και εταιρικής σχέσης πρέπει να συνδυαστούν με αυτή την επιτήρηση. Το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για τα Δημοκρατικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα καθώς και για την πυρηνική συνεργασία. Για διάφορους λόγους πολλές πάνε του κεφαλαίου 4, του τίτλου 4 δεν συζητιούνται από αυτή την οδηγία όπως οι δαπάνες για την κοινή πολιτική άμυνας την εξωτερική υπηρεσία, την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, τη μακροοικονομική βοήθεια και την ανθρωπιστική τη αυτή. Οι προτάσεις της Κομισιόν ζητούν την απλοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και μεγαλύτερη της ευελιξία που να επιτρέπει την ταχύτερη έγκριση τέτοιων αποφάσεων διότι πολλές φορές απαιτείται ταχεία πληρωμή ιδιαίτερα για ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις. Από απόψεις προϋπολογισμού πρώτον, η απλοποίηση. Ένας και μοναδικός κανονισμός θα απλοποιούσε τα πάντα και όλους τους τύπους βοήθειας που χορηγούνται. Θα ήθελα να τονίσω προς τους συναδέλφους και την Επιτροπή ΑΦΕΤ ότι αν εφαρμοστούν τεράστιες αλλαγές στον κανονισμό και υποκανονισμό, τότε θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται μια συνεπής στρατηγική για όλα τα εργαλεία. και να συνδυάζονται οι εξωτερικοί με τους εσωτερικούς μας στόχους ιδιαίτερα μέσω της απλοποίησης πρωτοβουλειών όπως τη στρατηγική 2020 δημοκρατία, ευνομία, ανθρώπινα δικαιώματα, επιχειρηματικό πνεύμα και προστασία του περιβάλλοντος. Και απ' την άλλη, αν ο κανονισμός θέλει να είναι καθολικής σημασίας, τότε πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά σε κάθε ένα μία από αυτές τις υπηρεσίες. Στα 6, 9 και 11 άρθρα γίνεται λόγος για εξαιρέσεις που δεν προσθέτουν τίποτα στην οριζοντιοποίηση ή την καθολικότητα του πλαισίου. Αναγνωρίζω ότι οι ιδιαιτερότητες της κάθε υπηρεσίας ή εργαλείου απαιτούν κάποιου ιδιαίτερους κανόνες περιορισμένου αριθμού, αλλά, αλλά λέγω, αυτό θα αναφέρεται στο κάθε συγκεκριμένο νομοθέτημα. Ο κανονισμός ο ίδιος πρέπει να διατηρεί τον καθολικό του χαρακτήρα και να περιορίζεται σε διαδικασίες πράγματι καθολικές για τη χρήση των δημοσιονομικών εργαλείων. Ο διαχωρισμός μερικών δράσεων σε δύο κανονισμούς δεν απλοποιεί τα πράγματα. Δεύτερον, η χρήση των αριθμών. Το 121 δισεκατομμύρια 8 προτείνονται να χορηγηθούν σε τέσσερις γεωγραφικές ενότητες και τρεις θεματικές. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 17,6% σε σταθερές τιμές. Άρα θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα ως προς τις εξωτερικές δράσεις θα ζητούσαν να χρησιμοποιούμε πάντοτε τέτοιες σταθερές τιμές διότι έτσι μπορούν να γίνουν πιο εύκολα συγκρίσεις, ιδιαίτερα μεταξύ πολιετών πλαισίων. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πιο μακρόπνο από ότι η ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού και πρέπει να καταλάβουμε ότι αν χρησιμοποιούμε τρέχουσες τιμές ε, δεν ε, πετυχαίνουμε το στόχο μας. Εκτός αυτού, δεν πρέπει να συζητάμε τα πράγματα μόνο βλέποντας το παρελθόν, αλλά να προβλέπουμε και εξελίξεις μακροοικονομικές και μακροχρόνιες, μακροπρόθεσμες. Μήπως προβλέπετε μελλοντική χρηματοδότηση περισσότερων χωρών. Ποια είναι η σχετική ανάπτυξη από περίοδο σε περίοδο κλπ. Ίσως η Κομισιόν να έχει τέτοιες προβλέψεις και αριθμούς, αλλά θα ήθελα αν έχει να τους καταστήσει επίσημους και να γίνουν γνωστοί και στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Γιατί είναι βασικό να έχουμε σωστούς αριθμούς, ιδίως γιατί εμείς ως κοινοβούλιο καμιά φορά κάνουμε πολύ εύκολα συμβιβασμούς και παραχωρήσεις. Τρίτον, οι κοινέ αξιολογήσεις. προτείνω η Κομισιόν στη μέση της περίοδου να μας γράφει μια έκθεση για όλες τις χρηματοδοτήσεις που επιτηρούνται, που αφορούν αυτό τον κανονισμό και ίσως και όλες τις εξωτερικές χρηματοδοτήσεις που να μην περιορίζονται μόνο στον τίτλο 4. να αναφέρεται γενικά το πεδίο εφαρμογής και χρήσης του κάθε κονδυλίου, ποιες ακριβώς είναι οι πληρωμές και οι συμμετοχές των εταίρων. Τέτοιου είδους εκθέσεις θα μας ήταν πολύ χρήσιμες ως αρχή συναρμόδια του προϋπολογισμού για να δούμε πού και πώς χρησιμοποιούνται τα ενωσιακά χρήματα και δεύτερον για να βελτιωθεί η ποιότητα της επιτήρησης και εποπτείας για μεγαλύτερη συνέπεια και συνδυασμό όλων των εργαλείων. Ένα παράδειγμα. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το εργαλείο, το ενταξιακό εργαλείο, από το μακροοικονομικό εργαλείο, από διαμεθοριακές χρηματοδοτήσεις κλπ. Και με από τη στρατηγική Τάνιουκ. Αλλά έτσι μπορεί και άλλες 100 χώρες να χρηματοδοτηθούν με παρόμοια εργαλεία και δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε όλα αυτά. Τέταρτον και όχι τρίτον. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του τι είναι κατεπίγουσα περίστασης και πρέπει να τους ενοποιήσουμε για να υπάρχει μεγαλύτερη νομική βεβαιότηση ως προς το αν και πότε πρέπει, αν μπορεί να αντιδράσει η Ένωση στην παγκόσμια κρίση. Πρέπει να αντιδρούμε μόνο σε περιστάσεις που όντως να είναι κατεπίγουσες για να απλοποιηθεί η λήψη αποφάσεων. Τέλος, το καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο δεν στοχεύει στην υποκατάσταση εθνικών εργαλείων ή ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ε, η Κομισιόν πρέπει να διασφαλίζει ότι ο χαρακτήρας χρηματοδότησής της θα είναι συμπληρωματικός με συνδυασμό τεχνογνωσίας και πληροφοριών από όλους τους ενδιαφερόμενους και τους εταίρους. Και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να μην επιβαρύνει άχρηστα την ε, δαπάνηση των υπολείπων ταμείων. Σας κατευχαριστώ. Merci, Madame le Rapporteur. Ε, Ευχαριστώ, εισηγήτρια. Κυρία Μονιός. Voilà, όχι Με Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Νέμσκι για την έκθεσή της. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και επειδή είναι και περίπλοκο αυτό το οριζόντιο μέσο, είναι κοινά τα στοιχεία από πολλά διαφορετικά μέσα και πολύ περίπλοκο το εγχείρημα να τα βρούμε. Συμφωνώ ε, ουσία με όλα σχεδόν από όσα είπατε, αλλά θέλω μερικές διευκρινήσεις για πολύ συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, οι οργανώσεις κοινωνίας πολιτών, ε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά αναφέρονται και στη σύντομη ε, αιτιολόγηση, αλλά και γενικότερα και στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και γίνεται λόγος για τη δυνατότητα για την ανάγκη διευκόλυνση συμμετοχής των οργανώσεων των, της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά αυτό αναφέρεται έτσι επιγραμματικά ε, στην αιτιολογική έκθεση, αλλά στο διατακτικό τίποτα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθεί και εκεί να κάνετε μια αναφορά στις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που είναι ερετά όργανα και επιλέξιμα μάλλον ε, για τη χρηματοδότηση. Σε ορισμένα από τα μέσα, ας πούμε στο μέσο γειτονία, αναφέρονται ερετά και στο προενταξιακό μέσο και κάπως συγκεχημένα και αόριστα στο μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, γι' αυτό νομίζω και στο οριζόντιο, μέσα στον οριζόντιο κανονισμό θα πρέπει να ε, υπάρχει μια τέτοια αναφορά. Δεύτερον, σωστά έχετε αναζητήσει ε, μια ισορροπία για τους στόχους της εσωτερικής πολιτικής και πώς θα ευθυγραμμιστούν ή θα συγκλίνουν με τους στόχους εξωτερικής πολιτικής για να είναι πιο Συνεπίσει οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία λοιπόν αναφέρεται η στρατηγική 2020, τη δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντο και πάει λέγοντα. Όλα αυτά είναι στοιχεία πάρα πολύ ευστοχά και ε, με εσωτερική και με εξωτερική διάσταση. Εκεί λοιπόν νομίζω θα πρέπει να αναφέρεται και τη μείωση της ένδυας γιατί εντάσσεται αυτό στη στρατηγική 2020 και σε κάποια άλλα μέσα που προσπαθεί να αναζητήσει κοινά στοιχεία τους η έκθεση. Σε σχέση με το μέσο δημοκρατίας και ανθρωπινών δικαιωμάτων, ορίζεται η δυνατότητα να χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το γραφείο του υπάτο ε, αρμοστού, της είπα της αρμοστίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς θα γίνει αυτό. Και με ποιε δαπάνε, πώς θα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την ύπατη αρμοστία ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λέτε στι τροπολογίες σα και είπατε και τώρα μόλι ότι διαφωνείτε με τις ειδικέ πρόνοιες ε, για κάθε ένα από τα μέσα αυτά σύμφωνα με τα άρθρα 6, 9, 10, 11. Τι εννοείτε ακριβώς. Κριτήρια επιλεξιμότητας είναι αυτά σε κάθε ένα από τα μέσα χρηματοδότησης για τις υποψηφιότητες. Πώς το λένε αυτό όταν υποβάλλουν υποψηφιότητα σε έναν διαγωνισμό. Για την πρόσκληση χρηματοδότησης των διαφόρων οργανώσεων στα διάφορα μέσα. Ακριβώς επειδή είναι διαφορετικά τα μέσα θα πρέπει να είναι διαφορετικές οι πρόνοιες και οι διατάξεις γιατί οι συνθήκες είναι διαφορετικές και οι ίδιες οι οργανώσεις μεταξύ τους. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι διαφορετικοί οι αποδέκτες και διαφορετικοί οι τρόποι υποβολής αίτησης και υποψηφιότητας για χρηματοδότηση. Αυτά. Κατά τα άλλα είναι πολύ σωστή και καλή η τρόπο η έκθεση γνώμη και θα κάνουμε τροπολογία στους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κυρία Μπραντνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Νέτσκι για τις καλές της προτάσεις. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά που είπατε εσείς για τη βελτίωση της εποπτείας. Εγώ έρχομαι εδώ από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που συζητήσαμε το μέσο για τη σταθερότητα όπου τα προγράμματα αυτοαξιολογούνται. Αυτό είναι λίγο αστείο. Όταν είσαι υπεύθυνο για ένα πρόγραμμα, για τη διαχείρισή του και σου ζητάνε να το αξιολογήσεις, ε, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα είναι τα καλύτερα. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εδώ σε επίπεδο συνοχής <clears throat> και συντονισμού και δεν θα πρέπει να δημιουργούμε επιπλέον επικαλύψεις ανάμεσα στα χρηματοδοτικά μέσα, γιατί κάθε μέσο μέχρι τώρα προσπαθεί από μόνο του να διευρύνει το πεδίο ε, που καλύπτει και αυτό δημιουργεί επιμέρους επικαλύψεις, κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ε, εμένοντας τη συνοχή και τον συντονισμό. Αναφερθήκατε επίση στον κατεπήγοντα χαρακτήρα της κρίσης. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν διαφορετικού κρίσεις. Οι κρίσεις καταρχάς που δεν μπορούμε εμείς να προβλέψουμε. Τυφώνες, πλημμύρες. Προβλέπονται από μία άποψη και πρέπει να αντιδράσει κανείς άμεσα. Και απ' την άλλη υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια και ό,τι χρειάζεται. Και απ' την άλλη υπάρχουν οι πολιτικές κρίσεις, οι οποίες πολλές φορές μπορεί κανείς να γνωρίζει από πριν α, τον εμφύλιο πόλεμο σε μια περιοχή. Τώρα θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα κατεπήγον πακέτο για τη Συρία σαν παράδειγμα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε πριν ένα χρόνο του τι θα συμβεί στη Συρία. Εν πάση περιπτώσει το θέμα αυτό είναι συνεχώς εξελισσόμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως ε, πολλές φορές περιορίζεται θα έλεγα στο όταν προσπαθεί να προβλέψει το τι θα συμβεί. Είμαστε πολύ κοντά στην ένοπλη σύραξη και καλό θα είναι να μπορεί κανείς να παρεμβαίνει σε πιο πρώιμο στάδιο, να υπάρχει ένα σύστημα προειδοποίησης όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά και αυτό θα είναι ευθυνότερο από ότι να παρεμβαίνουμε εκ των υξτέρων. Πολλές φορές βέβαια σε θέματα πρόληψης των συγκρούσεων των ενόπλων δεν υπάρχουν χρήματα γιατί δεν μπορεί κανείς να προβλέψει εύκολα. Αλλά πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο προβλεπτικοί και τουλάχιστον για τις πολιτικές κρίσεις να μην παρεμβαίνουμε μόνο όταν έχουν αρχίσει να πεθαίνουν πια οι άνθρωποι γιατί αυτό είναι ανεπαρκές. Κατά τα άλλα συμφωνώ με την κυρία Ευχαριστώ συνάδελφε. Η κυρία Τρούπελ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, αλλά το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξή. Στην έξι κυρία Σνέντσκι. Γιατί ήδη είναι ενταγμένο αυτό στο πρόγραμμα. Γι' αυτό είναι η βιωσιμότητα και η εφορία της εκπαίδευσης. 2% πηγαίνει στο λεγόμενο πρόγραμμα Εράσμους για όλους. Ανεξάρτητα από το αν θα διατηρηθεί αυτός ο τίτλος, είναι μια πολιτική ε, που ε, ενισχύει τις ευκαιρίες για τους νέους, τους δίνει καλύτερες ευκαιρίες να εκπαιδευτούν στους διάφορους τομείς και να σπουδάσουν. Και πραγματικά αυτό είναι επένδυση στο μέλλον. Και είναι σημαντικό στοιχείο του προενταξιακού μέσου και θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσαμε εκεί να κάνουμε περισσότερα. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ε, χώρες ε, ε, τις υποψήφιες έχουμε την ευκαιρία να προωθούμε την παιδεία και πολύ καλό είναι να συμπεριλαμβάνεται αυτό, αλλά ποτέ δεν θα φτάσουν τα λεφτά, είναι 2%. Ευχαριστώ. Merci, Elga. Ε, Χέλγα. Για να επανέλθω σε αυτό που έλεγε η κυρία Μπράντνερ, υπάρχουν και κρίσεις, περισσότερες είναι απρόβλεπτες και δράματα, άλλα που μπορούν να προβλεφθούν. Η κυρία Νέσκι, που έχει μεγάλη πείρα της εξωτερικής πολιτικής στη χώρα της, σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα της και για τα Βαλκάνια, θα μπορούσε να τα πει καλύτερα από μένα. Η τραγωδία της Ιουκοσλαβίας ήταν και προβλέψιμη και ε, ε, είχε προβλεφθεί και ε, το είχαν καταγγείλει. Έχουμε μέλη από τη Σλοβενία, παρατηρητές από την Κροατία και ελπίζω προσεχώς και άλλα μέλη από τις χώρες που προέκυψαν από την Ιουγκοσλαβική τραγωδία. Στο Σουδάν. Στο Σουδάν γνωρίζουμε και γνωρίζαμε ότι από τις 9 Ιουλίου του 2011 θα υπήρχε σοβαρή ε, απειλή πολέμου και μεγάλων ταραχών, γιατί ήταν η ημερομηνία που είχαν επιλέξει για μια διεθνή συμφωνία για ένα δημοψήφισμα που ξέραμε ότι θα κατέληγε σε απόφαση απόσχηση του Νοτιού Σουδάν από το Βόρειο. Και επίσης ευαισθήσαμε και την προσοχή της κυρίας Άστον μήνες πριν και στην Επιτροπή Εξωτερικών, αλλά και η δική μας Επιτροπή Προλογισμού για το κίνδυνο αυτό. Ε, πραγματικά εδώ είμαστε ασυγχώρητοι. Είναι αρκετές οι κρίσεις και τα γεγονότα που είναι τελείως απρόβλεπτα. Η ε, Αραβική Άνοιξη ουδής ε, μπορούσε να την προβλέψει, αλλά καμιά φορά γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος κρίσης κάπου. Υπάρχουν πράγματα που εξαρτώνται από τους διπλωμάτε την Επιτροπή Εξωτερικών και άλλα που εξαρτώνται από την Επιτροπή Προπολογισμών, έτσι ώστε να μπορούμε να κινητοποιούμε εγκαίρω τα μέσα και να έχουμε χρήματα με κάποια ευελιξία. Εξού και το πρόβλημα αυτό του κανονισμού για τις μεταφορές πιστώσεων και τις εκταμιεύσεις, έτσι ώστε να μην εμποδίζουν γραφειοκρατική φραγμή της επεμβάσης, όπως είπε η κυρία Μπράτμε μπορούμε να σώνουμε ζωές και να σταματούμε κρίσεις. Αλλιώς κοστίζουν οι κρίσεις αυτές και χρήματα αλλά και ανθρώπινες ζωές και πόνο. Κυρία Νέσχη, θέλετε να απαντήσετε και να παρουσιάσετε μια που θα έχετε και το λόγο και τη δεύτερη εκθεσή σας. Sorry, maybe just a few comments. Συγγνώμη, μερικά σχόλια απαντώντας στους συναδέλφους. Το πρώτο για την κοινωνία των πολιτών και το ρόλο της. Συμφωνώ πολύτος με τα όσα υπόθηκαν και θα καλωσόριζα οποιαδήποτε πρόταση για τα δικαιώματα, τα πολιτικά και τη φτώχεια. Πολύ σύντομα όντως θα πρέπει να ενταχθεί ε, παντού, αλλά αυτό είναι θέμα ε, της Επιτροπής Εξωτερικών, όχι του προπολογισμού και είναι και στην ατζέντα ε, την Ευρώπη 2020. Αλλά εμείς θα πρέπει κυρίως να επικεντρωθούμε τα δημοσιονομικά και τα υπόλοιπα στην Επιτροπή Εξωτερικών. Για τα άρθρα 6, 7, 8, 9 Διαφωνώ να συμπεριληφθούν στους γενικούς κανονισμούς. Μπορούν να γίνουν επιμέρους, ξεχωριστά στα διάφορα μέσα. Όχι στον κοινό κανονισμό. Τι άλλο. Παρακολούθηση. Μα γι' αυτό το λόγο προτείνω ενδιάμεση έκθεση με πληροφόρηση για τη χρηματοδότηση όλων των μέσων. Αυτό νομίζω μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Για τον κατεπήγοντα χαρακτήρα και πάλι. Συμφωνώ να είμαστε προσεκτικοί, αλλά πιστεύω ότι όταν έχουμε πολλαπλούς ορισμούς στα κείμενα, προκύπτουν συγχύσεις όταν πρόκειται για συγκεκριμένες διαδικασίες του προπολογισμού. Γι' αυτό θεώρησα σκόπιμο να το συμπεριλάβω στην πρότασή μου. Και τέλος, το εράσιμος για όλους. Ε, αυτό είναι το προενταξιακό μέσο, το IPA. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ε, χρησιμοποιείται παντού το πρόγραμμα αυτό παρά να έχω ένα ποσοστό στο κείμενο. Αυτά. Ως ε, απαντήσεις στα σχόλιά σας και στις ερωτήσεις σας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, να περάσω στην επόμενη έκθεση. Είναι γνωμοδότηση ουσιαστικά για το προενταξιακό μέσο Αυτός ο κανονισμός διέπει ένα μέσο, το μέσο της προενταξιακής βοήθειας, το IPA. Στη διατήρηση της κατάστασης στο σχεδιασμό και τους στόχους προγράμματος, ε, διατηρεί ως βασικό χρηματοδοτικό πυλώνα το IPA. 7,3% είναι η αύξηση με σταθερές τιμές στην περίοδο 2007-2013 για την επόμενη περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό ουσιαστικά θα δώσει μια ισορροπία ε, ανάμεσα στην πρόοδο για την επίτευξη των κριτηρίων ένταξης και θα βοηθήσει την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη στις δικαιούχες χώρες. Θα ήθελα εγώ να σας δείξω την πρακτική εφαρμογή άλλων ε, μέσων όπως είπα και προηγουμένως, για τον κοινό εφαρμοστικό κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για κάθε δικαιούχο χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής. Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε μία δικαιούχο χώρα για την περίοδο 2007-2013, με εξαίρεση την Κροατία, θα κυμαίνεται μεταξύ 10 και 30% στο τέλος της περίοδου. Παρόλο που η κατακεφαλή χρηματοδότηση θα μπορούσε να αποτελεί αξιόπιστο δίκτυ για διάφορους λόγους, πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε τους λεγόμενους μακροδείκτες που μετρούν τη συνολική στήριξη σε σύγκριση με το ΕΠ κάθε δικαιούχου χώρας, έτσι ώστε να αποτυπωθεί πλήρως η προστιθέμενη αξία και τα καθοριστικά θετικά εξωτερικά στοιχεία της ενωσιακής χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, Καθώς οι δικαιούχες χώρες δημιουργούν και τελειοποιούν τις απαραίτητες οικουμενικές αρχές που αποτελούν ισχυρές κινητήρες δύναμης της οικονομικής ευεξίας, μπορεί να φαίνεται λογικό να αλλάξουμε την εστίαση από τις κατακεφαλήν ποσότητες σε μικρούς δείκτες, ώστε να αποτυπωθούν οι συστημικές και ποιοτικές αλλαγές. Κατά συνέπεια, αριθμητικά, σε πραγματικούς όρους η αύξηση θα πρέπει ε, να είναι όχι μικρότερη από τη σωρευτική πραγματική αύξηση του ΑΕΠ. Ο αριθμός των χωρών με πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το μελλοντικό μηχανισμό μειώνεται σε 8 λόγω της ένταξης της Κροατίας, κάτι το οποίο ενδεχομένως μεταβάλλει τη συγκριτική κατανομή εντός του συνόλου της χρηματοδότησης και από την οπτική γωνιά των δικαιούχων ευνοεί την πρόσβασή τους στις πιστώσεις αν θέλουμε να δούμε ακριβώς τα στοιχεία τα αριθμητικά τα οποία προέρχονται από τη χρήση των ποσών αυτών χωρίς εξαιρέσεις εκτός βέβαια από την Κροασία από την Κροατία συγγνώμη, η πραγματική αύξηση των πιστώσεων από τη μία περίοδο στην άλλη θα πλησιάζει το 20%. Μάλιστα με τις προτινόμενες αλλαγές όλες οι χώρες που δικαιούνται πρόσβαση στη χρηματοδότηση θα εστιάζονται στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη που μέχρι τώρα ήταν απρόσιτες, ιδιαίτερα για τις υποψήφιες χώρες. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό για χρηματοδότηση στις χώρες που χρησιμοποιούν τους τομείς αυτούς και αυτό ίσως να δημιουργήσει και περισσότερο ανταγωνισμό για χρηματοδότηση στους ίδιους τομείς και ίσως να αλλάξει πιθανόν και το επίπεδο πρόσβασης ορισμένων αποδεκτών σε αυτές τις πιστώσεις. Επιπλέον τούτου και επιπλέον ακριβώς των βελτιωμένων διοικητικών δυνατοτήτων των αποδεκτών μετά από το IBA 1 ή MIPV 1 οι χώρες αυτές θα οδηγηθούν σε μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης κεφαλαίων και προεφοδιασμού κατά τα πρώτα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κανείς από την πρόσβαση στους κοινοτικούς πόρους και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν προετοιμάζουμε και τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Να πω ότι αυτές οι εξελίξεις δεν ε, αποκλείουν κανένα από δίκαιη πρόσβαση ε, λόγω ακριβώς της μείωσης των ενωσιακών πόρων, ιδιαίτερα στον τομέα της οικοδόμησης θεσμών. Να πω επίσης ότι υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία στην πρόταση. Τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή αποσκοπούν στο να καταστήσουν τους πόρους πιο ορθολογικούς και ευέλικτους. Ναι. Υπάρχουν ορισμένες πλευρές οι ναι. οποίες δεν αντιμετωπίζονται με τον σωστό τρόπο και μας δημιουργούν ανησυχίες. Πρώτον, το αποθεματικό επίδοσης όπως λέει η αιτιολογική έκθεση, το αποθεματικό επίδοσης θα είναι ευπρόσδεκτο και θα είναι ένα κίνητρο για επιδόσεις. Παρ' όλα αυτά δεν παρουσιάζεται νομοθετικό κείμενο γύρω από την ιδέα αυτή. Εγώ κάνω την πρόταση αυτή, λέγοντας ότι αυτό το αποθεματικό θα πρέπει να δημιουργηθεί υπό τον πλήρη έλεγχο της αρχής του προϋπολογισμού, με εμπλοκή ικανοποιητική του Κοινοβουλίου και παρακίνηση προόδου στις αποδέκτριες χώρες. Οι τομεακές στηρίξεις θα μπορούν να βασίζονται σε συγκεκριμένους δείκτες, αν και αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία της γενικής δημοσιονομικής στήριξης δεν προσμετράται εύκολα. Το δεύτερο είναι ο εξορθολογισμός των στόχων των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να συνδέεται με την πολιτική διεύρυνση έτσι ώστε να δημιουργούνται μακροπρόθεσμα αμοιβαία και αυτοανισχυόμενα ωφέλη. Θα ήθελα να προτείνω οι στόχοι του εξορθολογισμού να έχουν ε, καθοριστική παρουσία στους στόχους του προγράμματος Ευρώπη 2020, ενσωμάτωση δημοκρατίας, κράτος δικαίου, περιβάλλον κτλ. Και τέλος, οι στόχοι και τα κριτήρια. Θα ήθελα να πω ότι οι ορισμοί των στόχων και των κριτηρίων για την βοήθεια αυτή θα πρέπει να υπακούν συγκεκριμένους ξεκάθαρους δείκτες. Πέραν από τους δείκτες που προτείνονται στο ψήφισμα θα ήθελα να προτείνω να προσθέσουμε και νέες δυνατότητες δημοσιονομικής σταθερότητας, φορολογικής σταθερότητας και άλλων κριτηρίων στο σύνολο των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται. Τέλος, η μεγαλύτερη συνοχή. Απαιτείται η διασφάλιση μεγαλύτερη συνοχή συντονισμού και απαιτούνται και συνεργίες ανάμεσα στις διαθέσιμες εσωτερικές και εξωτερικές χρηματοδοτήσεις για τους δικαιούχους. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τα πλεονεκτήματα τα οποία προέρχονται από την χρηματοπιστωτική μόχλευση, κάτι το οποίο θα μεγιστοποιήσει τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων αυτών από τα ποσά τα οποία θα διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πιστοτικά ιδρύματα. Αναγνωρίζουμε όμως ότι η χρήση των ευρωπαϊκών πιστώσεων θα πρέπει να σέβεται τους βέλτιστους κανόνες όπως προβλέπουν οι δημοσιονομικοί κανονισμοί και οι εφαρμαστικοί κανονισμού. Το πλαίσιο επένδυση στα Δυτικά Βαλκάνια ήταν μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση, συνδυασμό και απόδοση σε μέτρα στήριξη σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα ήθελα να πω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στον διάλογο για την βοήθεια, το συντονισμό της βοήθειας υπό το πνεύμα ακριβώς του πλαισίου ενίσχυσης των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ ε, την κυρία Νέσκη ο κύριος Φέρμα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, ευχαριστώ την Επιτροπή. Οι προτάσεις για το πρόγραμμα αυτό ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση και από την Επιτροπή και από την εισηγήτρια. Κάποια θέματα όμως πρέπει να συζητηθούν περισσότερο και εδώ θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες Έχουμε και κάποιες, ε, θα έλεγα, φρέσκες εντυπώσεις ε, μετά από την αντιπροσωπεία που κάναμε στην Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα υπό την Προεδρία του κυρίου Ντεχάν και νομίζω ότι θέματα που γνωρίσαμε εκεί θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Καταρχάς, το νέο πρόγραμμα είπα θα πρέπει να πιο ευέλικτο. Τώρα έχει επτά διαφορετικά κλάδους θα έλεγα, οι οποίοι είναι κάπως δίσκαμπτοι. Πρέπει να καταλήξουμε σε λύσεις πιο ευέλικτες και πιο αποτελεσματικές. Όταν λέμε αποτελεσματικές δεν το λέμε μόνο για τους χρήστες, θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και για την Ένωση η παρέμβαση αυτή. Η απλούστευση είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα έλεγα έχει πολύ μεγάλη σημασία σαν παράδειγμα η χρηματοδότηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών, η χρηματοδότηση ε, των ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών επιτόπου κτλ. Τώρα κάποια επιπλέον συγκεκριμένα σημεία. Συντονισμός των δωρητριών χωρών και οργανισμών. Ένας πίνακα συνεργασίας ανάμεσα στον πίνακα ΙΠΑ, στα κράτη-μέλη που μερικές φορές χρηματοδοτούν άμεσα κάποια προγράμματα θα πρέπει να βρούμε τρόπους εν πάση περιπτώσει για να αποφύγουμε και κενά αλλά και επικαλύψεις, γιατί και τα δύο υπάρχουν σήμερα. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξουν κάποιες σωστές διατυπώσεις από πλευράς της εισηγητρίας. Να υπάρξουν και κάποιες επιπλέον τροπολογίες γύρω από τα θέματα αυτά για τη σημασία του διαλόγου ανάμεσα στις δωρήτριες χώρες και υπηρεσίες και οργανισμούς μάλλον, γιατί αλλιώς διατρέχουμε τον κίνδυνο να φανούμε αναποτελεσματικοί. Δεύτερον, η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητάμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Τουρκία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που την χάνει ενίσχυσης. Είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τις τοπικές δυνατότητες, τις περιφερειακές δυνατότητες και για τους κοινωνικούς εταίρους και για την αγορά εργασίας και για την κοινωνία των πολιτών. Συναντηθήκαμε με πολλούς από αυτούς στην Τουρκία και εδώ έχουμε τεράστιες διαφορές ανάμεσα βέβαια σε αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία και στις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στις οποίες δεν υπάρχει η δομή, η διάρθρωση για τις δυνατότητες βελτίωσης της παρέμβασης της κοινωνίας των πολιτών. Ταυτόχρονα η χρηματοδότηση, αν θέλετε, της κοινωνίας των πολιτών μοιάζει με τα ψίχουλα που τους δίνουμε όταν έχουν δοθεί τα χρήματα αλλού και παίρνουν ό,τι περισσέψει. Πρέπει αυτό σαν αντίληψη να αλλάξει. Υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες αναφέρονται και κάνουν προτάσεις για συγκεκριμένα ποσοστά του ταμείων αυτών που θα πρέπει να πηγαίνουν στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό το σκεφτούμε αυτό. Πάντως είναι θέμα να προσπαθήσουμε να διασώσουμε την αυτονομία αυτών των μέσων. Τώρα, για τα χρηματοδοτικά μέσα και χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν είναι δυνατόν ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να χρηματοδοτεί ό,τι ακριβώς εμείς επιθυμούμε, τα πάντα. Υπάρχουν ανάγκες και για υποδομές και για βαριές επενδύσεις, αλλά και για κάποιες ίσονες παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν την κοινωνία των πολιτών. Απαιτούνται επιπλέον χρηματοδοτικά μέσα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Πέραν αυτών δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφωνία. Πρέπει να υπάρχει επίσης και μια κοινωνική διάσταση στον κανονισμό ΙΠΑ. Αν μιλάμε για τη στρατηγική 2020, Ευρώπη 2020, να μην ξεχνάμε ότι η στρατηγική αυτή δεν αφορά μόνο τις ε, ε, συγκεκριμένες παρεμβάσεις και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και μια σημαντική κοινωνική διάσταση. Βλέπουμε ποιες χώρες την χάνουν ενίσχυση, η Τουρκία σαν παράδειγμα. Ένα από τα προβλήματά τους δεν είναι η ρυθμή ανάπτυξης, γιατί το, δεύτερο, το επίπεδο ανάπτυξης Τουρκίας είναι το δεύτερο καλύτερο στον κόσμο μετά από την Κίνα. Το πρόβλημα είναι οι τεράστιες διαφορές οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στις κοινωνικές κατηγορίες, εκ των οποίων κάποιες αναπτύσσονται και κάποιες όχι. Λοιπόν, η κοινωνική διάσταση είναι απαραίτητη, απαραίτητη να καλύψει ιδιαίτερα τις ε, λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Πέμπτον είναι η δημοσιονομική στήριξη. Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις για τη δημοσιονομική στήριξη, κάτι το οποίο απαιτεί λιγότερες διοικητικές ε, ε, ε, παρεμβάσεις. Θα πρέπει να μην αγνοούμε εδώ ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από ισχυρά μέτρα καταπολέμησης της διαφοράς. Mm. Είναι απαραίτητη η καταπολέμηση της διαφθοράς και όχι ο περιορισμός στην δημοσιονομική ενίσχυση. Η κυρία Νέινσκι επίσης αναφέρθηκε σε, πολλά τεχνικά, σε πολλές τεχνικές και ε, οικονομικές προϋποθέσεις. Ερεσιμότητα, ε, αυτή που είπαμε το αποθεματικό επιδόσεων, τέτοια πράγματα τα οποία όταν συζητούσαμε με τους φίλους μας στην Τουρκία μας έλογαν ε, ότι μας αδικείται γιατί κατά κεφαλήν εμείς παίρνουμε πολύ λιγότερα από ό,τι άλλες χώρες. Βέβαια η Τουρκία είναι 10 φορές μεγαλύτερη από τις άλλες χώρες τουλάχιστον. Οπότε ε, μια τέτοια χώρα επηρεάζει θα έλεγα τα ποσά που έχουμε στη διάθεσή μας με τρομερό τρόπο. Δεν μπορούμε να δίνουμε λοιπόν ενισχύσεις στις χώρες αυτές επί τη βάση της, ε, του δίκτυ θα έλεγα του πληθυσμιακού αυστηρά. Τώρα, ε, για τα ίδια προβλήματα έχουμε και για τα δικά μας, αν θέλετε, τα μία συνοχής. Το θέμα δηλαδή της αιρεσιμότητας, το θέμα της, του αποθεματικού επιδόσεων κτλ. Εδώ μπορεί να έχουμε διαφορές, γιατί μπορεί σαν παράδειγμα να μην συμφωνήσουμε με τη λεγόμενη μακροοικονομική αιρεσιμότητα την οποία προτείνει η κυρία Νάισκε. Για πάρα πολλά χρόνια έχουμε προπαρασκευαστικές δράσεις στον τομέα της αποκατάστασης πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές ενόπλων συγκρούσεων. Έχει πάρα πολύ σημασία εδώ ε, να προχωρήσουμε με τέτοιου είδους προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά προγράμματα που ήταν επιτυχή στο παρελθόν. Θα πρέπει να υπάρξει πλέον συγκεκριμένη αναφορά σε τέτοιου είδους προγράμματα, ιδιαίτερα σε περιοχές σύγκρουσης διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η προσπάθεια αυτή για τη συμφιλίωση διαφορετικών ομάδων. Να αποδείξει κανείς ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια χρήματα για την ανοικοδόμηση μιας εκκλησίας και την ανοικοδόμηση ενός τεμένου στη Βοσνία, αυτό είναι κρίσιμο για την προσπάθεια ανοικοδόμησης της χώρας. Απαιτείται λοιπόν εμείς να συμπεριλάβουμε κάποιες συγκεκριμένες αναφορές στο θέμα αυτό της αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομίας στο μέλλον. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Θα καταθέσουμε αρκετέ τροπολογίε. οι περισσότερε δεν θα είναι θα έλεγα αμφισβητήσιμε. κάποιες οι οποίε αφορούν την μελλοντική μακροοικονομική αιρεσιμότητα παρουσιάζουν κάποια θέματα. Ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφοι. Ο κύριο Κόβατ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα καλωσορίζω εδώ στην πρώτη σας συνεδρίαση. Πρόκειται για παρατηρητή από την Κροατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω μερικά λόγια με βάση την κροατική εμπειρία και σε σχέση με την τη διαμεθοριακή συνεργασία και τον έρασμο για όλους και όλες. Η απλοποίηση είναι κάτι πολύ ωραίο από πολλές απόψεις όχι μόνο για τις ΜΚΙ όμικρον, αλλά και για τοπικές κοινότητες και δήμους που σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν μπορούν καν να αιτηθούν για χρηματοδότηση το ίδιο μπορούμε να αναμένουμε ότι ισχύει και στη Βοσνία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη. Πρέπει να δούμε πώς μπορούν να απλοποιηθούν όλα αυτά και να αλλάξουν ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες, τέτοιες συνθήκες, ώστε όσοι χρειάζονται περισσότερο τα προγράμματα να μπορούν να χρηματοδοτούνται. Δεύτερον, η διαμεθοριακή συνεργασία που μπορεί να σχετίζεται και με το πρώτο θέμα που ανέφερα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την συμφιλίωση εθνών που μπορεί στη δεκαετία του 90 και στις αρχές και ακόμη και του 2000 να είχαν μπλακεί σε σειράξεις. Οι παραμεθόριες περιοχές αυτών των χωρών είναι πάντοτε υπανάπτυκτες και γι' αυτό στηρίζουμε όλα τα προγράμματα διαμεθοριακής συνεργασίας ως σημαντικό στοιχείο του ΙΠΑ ιδίως στις χώρες της πρώην Νοτιοσλαβίας. Όσο δε για τη βιωσιμότητα της παιδείας Εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεπ και βλέπω ότι η βιωσιμότητα της παιδείας από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο χειροτερεύει από χρόνο σε χρόνο και η ποιότης αλλά και η προσβασιμότητα στην παιδεία κινδυνεύουν Δέχομαι λοιπόν αυτή την πρόταση του 2% για τον έρασμο για όλους και όλες. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε ή δυνατόν να αυξηθεί το ποσοστό αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ μου συνάδελφε. Η κυρία Νίμσκι θέλει μήπως να ξανααπαντήσει εκ νέου. Ναι, πολύ σύντομα όμως. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Γκουέρμ για τη σημαντική γνωμοδότηση και για τα σχόλια. Έχουμε γνωμοδότηση και για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τη διεύρυνση. Γι' αυτό χαίρομαι πολύ για αυτά που είπε. όταν ψηφίσουμε θα λάβουμε υπόψη αυτά που είπατε. Και ευχαριστώ και τον Κροάτη συνάδελφο διότι τα περισσότερα από αυτά που ανέφερε τα ξέρω και εγώ από δική μου εμπειρία και στηρίζω απόλυτα αυτά που είπε. Η απλοποίηση, η διαμεθοριακή συνεργασία είναι πολύ σημαντικά πράγματα για την βιωσιμότητα του εκδημοκρατισμού στα Δυτικά Μπαλκάνια. Ευχαριστώ πολύ τους πάντες και τις πάσες. Ευχαριστούμε πολύ κυρία εισηγήτρια. Και για τις δύο αυτές εκθέσεις έχουμε το ίδιο ημερολόγιο χρονοδιάγραμμα. 22 Μαΐου λίγη η διορία κατάθεση τροπολογιών. Ετοιμάστε τροπολογίες λοιπόν. Η έκθεση θα εγκριθεί στις 20 και 21 Ιουνίου για να ε, ψηφιστεί στην ΑΦΕΤ τον Ιούλιο στην ΑΠΕΞ και φαντάζομαι ότι μετά τις διακοπές θα, περάσει στην θα περάσουν στην Ολομέλεια. Ωραία, τώρα τηρήσαμε πλήρως το προτινόμενο χρονοδιαγραμμά μας και τώρα θα ψηφίσουμε voting time και μετά θα, θα εξετάσουμε την έκθεση Ριβελίνη μαζί με τους συναδέλφους της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού που θα έρθουν να καθίσουν εδώ δίπλα μου σε λίγο. Λοιπόν, το σημείο 14 έχουν ζητηθεί και δύο αιτήσει μεταφοράς στον προϋπολογισμό του 12 η Φραντσέσκα Μπαλτζάνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση περίθμου 3, όπως προβλέπεται από το δημοσιονομικό κανονισμό, προτείνει την χρήση ένα ποσό 120.000 ευρώ από το Ταμείο Προσαρμογής για να δοθεί τεχνική βοήθεια στις χώρες μέλη για τη χρήση του Ταμείου. Είμαστε κάτω από το ελάχιστο ποσό για τη χρήση που είναι το 0,35%. Συνεπώς η πρότασή μου είναι να υπερψηφιστεί ακριβώς αυτού του είδους η επιστροφή. Αντίθετα για την επιστροφή 5 αφορά το αποθεματικό το οποίο είχαμε ψηφίσει στον προϋπολογισμό του 2012 για την επιτροπολογία και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Εγώ είχα βάλει μια επιφύλαξη στα ποσά αυτά, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μεγαλύτερες προσπάθειες έτσι ώστε να μας ξεκαθαρίσει το αίτημά της και να μπορέσουμε εμείς να νερέσουμε την επιφύλαξη. Έχω λοιπόν επιφύλαξη κατά τις 5. Très bien, je vous remercie. Alors, on va d'abord examiner le 3. Καλώς, θα εξετάσουμε το 3 πρώτα. Έχεις δει το λόγο και ο Σάλβαρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά τη συνάδελφο Μπαζάνη. Τι μας είπε για τη μεταφορά πιστώσεων. Γιατί εμείς θα προτείναμε απόρριψη γιατί δεν έχει ψηφιστεί η έκθεση. Αυτό είπε η κυρία Μπαζάνη. Συγγνώμη γιατί περιτεύει τότε η δική μου τοποθέτηση. Δεν κατάλαβα τι μας είπε. Όχι, κοιτάξτε λέει ο Πρόεδρος, υπάρχουν δύο διαφορετικές μεταφορές, δύο διαφορετικές πιστώσεις. Κυρία Μπαλτζάνη, παρακαλώ να επαναλάβετε, γιατί ο κύριος Σάλβαρο προφανώς δεν σας κατάλαβε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, υπάρχουν δύο οι επιστροφές που προβλέπονται εδώ, η παρίθμου 3 και η παρίθμου 5. Προτείνω να υπερψηφιστεί το 3. Αυτό αφορά την χρήση ενός ποσού από το Ταμείο Προσαρμογής, ένα μικρό ποσό ουσιαστικά, για την τεχνική βοήθεια προς τα κράτη-μέλη, για τη χρήση ακριβώς του ιδίου του Ταμείου. Σας ζητώ λοιπόν να υπερψηφίσετε τη συγκεκριμένη αυτή επιστροφή. Τώρα το 5 αφορά την απόσυρση μιας επιφύλαξης την οποία εμείς είχαμε θέσει σε μια γραμμή του προϋπολογισμού σχετική με την επιτροπολογία και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Αυτά τα είχαμε βάλει στο αποθεματικό λέγοντας ότι σαν κοινοβούλιο εμείς θα αλλάζαμε την άποψή μας αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδινε καλύτερες διευκρινήσεις για το ρόλο αυτών των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Δεν μας δόθηκαν τέτοιες εξηγήσει και γι' αυτό προτείνω να καταψηφίσουμε την πρόταση 5 περιμένοντας περαιτέρω εξηγήσει και διευκρινήσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, συνάδελφοι, καταλάβατε. Α, σωστά κατάλαβα τότε και με καθησυχάζει γιατί μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι τουλάχιστον την τρία θα την καταψηφίσουμε. Υπάρχει η έκθεση για τη μεταφορά πιστώσεων, αλλά δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή. Δηλαδή πώς θα κάνουμε μεταφορά πιστώσεων χωρίς να έχει εγκριθεί η αντίστοιχη έκθεση. Αυτό το θέτω στην κρίση της εισηγήτριας. Το θεωρώ λάθος να το υπερψηφίσουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε την εξή δυσκολία την οποία θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να είχαμε αποφύγει. Να εγκρίνουμε πρώτα τη νομική βάση και μετά τη μεταφορά πιστώσεων. Ωραία. Η νομική ε, βάση είναι στην έκθεση του κ. Κοσλόφσκη και δεν μπορούμε σήμερα να την εγκρίνουμε. Μπορούμε να μην ψηφίσουμε τη μεταφορά πιστώσεων αν θέλετε, αλλά πιέζει ο χρόνο, λίγη προθεσμία. Και στη συνέχεια η σιωπή μας ε, θεωρείται συνένεση και λίγη την πέμπτη η προθεσμία. Τώρα είναι θέμα αρχής και επιλογή. Η Επιτροπή Προπολογισμών θέλει να εκφραστεί. Αν θέλει, αν υπάρχει πλειοψηφία, ότι είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής. Για την ίδια τη χρηματοδότηση και την αρχή για το πρόγραμμα τεχνικής ε, βοήθειας, το συζητήσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Κοσλόφσκι, είναι μεγάλη συνένεση, οπότε και ψηφίζουμε. Άλλος, χάνουμε την προθεσμία και έτσι κι αλλιώς, ε, εφόσον δεν θα έχουμε διαφωνήσει, η σιωπή θα εκλειφθεί ως θετική γνωμοδότηση Επιτροπής Προπολογισμών. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι ούτως ή άλλως και προφανώς οι πιστώσεις δεν θα μπορέσουν να καταβληθούν, οι πληρωμές δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο όταν θα έχει εγκριθεί νομική βάση. Έτσι έχει το πρόβλημα. Η συγκήτριά μας είναι υπέρ της μεταφοράς πιστός. Παρά αυτό το λάθος χρονοδιάγραμμα και για το οποίο εμείς ευθυνόμαστε. Θα φροντίσω το μέλλον να μην επαναληφθεί. Δεν είναι απολύτως ευχάριστη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, να ψηφίσουμε με τη σειρά. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς πιστώσεων παρελθόν 3. Ευχαριστώ. Κατά. 3, 4, 5, 6, 7, 7. Bien, abstention. Εποχές. Εγκρίνεται τη μεταφορά αυτή. Παριθμό 3. Καλώς. Για την 5 όμως, δηλαδή την ε, άρση του αποθεματικού διαφωνεί η συγγητρία. Υπέρ. Μερικοί κατά. Όλοι. Ομόφωνα σχεδόν. Απορρίπτεται η μεταφορά και διατηρούμε το αποθεματικό. Θεωρεί η συγγήτρια ότι δεν έχουμε ακόμα επαρκείς πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε αρκετά καθυσυχαστικές. Σας ευχαριστώ. Για τα άλλα θεσμικά όργανα δεν υπάρχει αίτημα μεταφοράς πιστώσεων και περνούμε στο σημείο 16 της Μόνικα Χολμάγερ. Πολιτική ακινήτων. Μας προτείνετε να λάβουμε απόφαση, κυρία Χολμάγερ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, μάλιστα. Θα ήθελα να σας κάνω μία πρόταση, αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ähm, Ξέρετε ότι ε, είναι μεγάλη ιστορία αυτού του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και πολύ υπαρθή στο Κοινοβούλιο και θα σας παρακαλούσα Πρόεδρε αφού έχουμε τα έγγραφα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ καλά και πολύ ενδιαφέροντα αλλά είναι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής όλα αυτά. Ε, το ύψος του κόστους ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Ακόμα δεν έχουμε ούτε τους διαγωνισμούς ούτε τίποτα. Και έχουμε μερικές ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε τη μορφή γνωμοδότησης τέλη Μαΐου. Γι' αυτό θα παρακαλούσα σήμερα να αποφασίσουμε ότι θα γνωμοδοτήσουμε και το έχω συζητήσει με τους συνεισηγητές που αισθάνονται και αυτοί σαν εμένα να κάνουμε γνωμοδότηση γιατί βέβαια αυτό το έργο θα θέλαμε να το παρακολουθήσουμε σωστά, να το συνοδεύσουμε όπως ε, αρμόζει και σήμερα θα παρακαλούσα να αποφασίσουμε ότι θα κάνουμε γνωμοδότηση και όχι μεθαύριο. <laughs> Δηλαδή θέλω να έχω λίγο χρόνο να το συζητήσω με τους εισηγητές. Δηλαδή τέλη Μαΐου θα προτείναμε, όχι την επόμενη συνεδρίαση αλλά τη μεθεπόμενη για την γνωμοδότηση. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, μας συμβουλεύετε να γνωμοδοτήσουμε. Όχι αυτή τη βδομάδα λοιπόν, αλλά τέλη Μαΐου, στην επόμενη φορά. Έχουν ζητήσει δύο το λόγο. Πρώτος ο George Λάιον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω την πρόταση της Μόνικα να γνωμοδοτήσουμε για αυτό το έργο μετά την επίσκεψη στο κτίριο ΚΑΤ στο Λουξεμβούργο, βγήκαν στην επιφάνεια διάφορα ανησυχητικά ως προς τη διαχείριση των έργων και τη δυνατότητα των αρχών του Κοινοβουλίου να ολοκληρώνονται τα έργα ε, εγκαίρως και στη συμπεφωνημένη τιμή. Βγήκαν στην επιφάνεια διάφορα πράγματα που ανησυχούν την Επιτροπή μας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κτίριο, είναι νωρίς ακόμα, είναι το στάδιο της ε, προκήρυξης διαγωνισμού. Βεβαίως θα κοιτάμε θέματα προπολογισμού ε, και την επίπτωση στον προπολογισμό. Δεν θα διαχειριστούμε το project ή το κτίριο, αλλά θα πρέπει ε, να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματά μας θα πιάσουν τόπο και θα συνοδεύσουμε το έργο αυτό έτσι ώστε να οδηγηθεί σε αίσιο πέρας και με επιτυχία να ολοκληρωθεί γιατί έτσι και λιώς επικρίσεις θα δεχθούμε ό,τι και να κάνουμε. Ελπίζω να συμφωνήσει και η Επιτροπή, να γίνει γνωμοδότηση και η Επιτροπή Προπολογισμού να συνδεθεί σε αυτή την προσπάθεια. Και να συμμετέχει πάρα πολύ υπό τη δημοσιονομική όμως ε, επιτυχή. Να βεβαιωθούμε ότι γίνεται σωστή και χρηστή διαχείριση. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Η κυρία Μπέρζο Μωράτα. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι Σκιώδη συγγήτρια εξ ονόματος της ομάδας μου και θα ήθελα να πω ότι σε περιόδους δημοσιονομικών περικοπών στα κράτη-μέλη θα πρέπει ξανά και ξανά να εξετάζουμε την κάθε μας ε, επένδυση και χαίρομαι που μαζί της γνωμοδότηση. Συμφωνώ με την ιδέα του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, αλλά θα πρέπει να γίνεται και έρευνα εκεί, όχι μόνο πληροφόρηση ε, στους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχουν μερικά θέματα που συνδέονται με αυτό. Ε, η ε, μετασκευή του κτηρίου χρειάζονται έργα. Θα πρέπει να απομακρυνθεί ο αμίαντος, να διευρυνθεί το κτίριο, να επεκταθεί και να γίνουν κάποια έργα επισκευής. Χρειάζονται και μελέτες. Δεν ξέρω, έχουν ε, κατατεθεί μελέτες αυτές ήδη για να αποφασίσουμε αν χρειάζεται επέκταση του κτηρίου ή απλή ε, μετασκευή του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα πρέπει να συνεργαστεί και με άλλα θεσμικά όργανα για τη χρηματοδότηση. Έχει δεσμευτεί, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Και σας παραπέμπω στην έκθεσή μας για τον προπολογισμό του 2012. Καλωσορίσαμε τις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα συμμετέχει και θα υποστηρίξει αυτό το έργο. και πιστεύω ότι ο όγκος ευρωπαϊκής ιστορίας είναι ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο και η Επιτροπή μας καλό θα είναι να έχει και γραπτή νομοδότηση και συμφωνώ. Ο κύριος Χάρτουγκ. Πρόεδρε, χαίρομαι με την πρόταση της κυρίας Χολμάιερ για γνωμοδότηση από πλευράς Επιτροπής μας και καλό θα ήταν να γράψουμε στη γνωμοδότηση ε, αλλά ε, ε, δεδομένου του παρόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σκόπιμο τώρα να κάνουμε ένα οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας για το παρελθόν. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Υπάρχει ήδη τοποθέτηση όντως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή στο κόστος και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο διάκειται θετικά και είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει. Από πλευρά μα ήταν έτσι κι αλλιώ προαπαιτούμενο, γιατί το θέμα του οίκου τη Ευρωπαϊκή Ιστορία δεν είναι απλώ ε, θέμα του Κοινοβουλίου, είναι ιδιαίτερη παρουσίαση τη μεταπολεμική ιστορία, πώ δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στη συνέχεια η Ένωση και όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την ιστορία τη. Και βεβαίω είναι και η ιστορία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή και όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει δηλώσει ότι θα συμμετέχει, θετικά λοιπόν απάντησε και χαίρομαι ε, που συμφωνεί ο κύριος Χάρτον για τη γνωμοδότηση, αλλά μάλλον θα είναι διαφορετική η γνώμη μας τελικά για το εάν χρειάζεται να δημιουργηθεί ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ως εισηγήτρια θα κάνω μεγάλη συζητήσεις με τους συναδέλφους που αποφάσισαν να γίνει αυτό το έργο, αλλά θα πρέπει να γίνει με, σύνεση, με λογική, με παρακολούθηση και από πλευρά μα. Γι' αυτό το επόμενο διάστημα παραμένουν πολλά ερωτήματα ανοιχτά και θέλουμε να τα πούμε έτσι στεναρά και στη γνωμοδότησή μας, έτσι ώστε να συνοδεύουμε τη φάση αυτή τώρα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης και της προκήρυξης από την αρχή. Γενικά η πολιτική ακινήτων του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου είναι κάτι που αφορά άμεσα τους βουλευτές και θα πρέπει να είναι πάντα πολύ καλά ενημερωμένοι ε, και έτσι κι είναι μια πάγια συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα σας παρακαλούσα να πάρουμε αυτή την απόφαση για γνωμοδότηση. Très bien. Je σας ευχαριστώ. Συμφωνούν όλοι λοιπόν με την εισηγήτρια για αυτά τα δύο σημαντικά θέματα. Πρέπει να γνωμοδοτήσουμε και να έχουμε αρκετό χρόνο. Δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε ούτε σήμερα ούτε την επόμενη Πέμπτη. Στην επόμενη συνεδρίασή είμαστε τρει τρεις Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Κάναμε όλες τις ψηφοφορίες και τώρα το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Όχι, όχι. Α, ε, τότε συγγνώμη. Ορίστε Μόνικα. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Έχω και δεύτερο θέμα. Το κτίριο Σιάνς ΑΓΕ, Συνοδόμων του ΑΓΕ 30, όπως γνωρίζουμε το κτίριο Ίστμαν είναι σε σχετικά κακή κατάσταση. Οπότε, ανεξάρτητα από τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας, έτσι και αλλιώς εκείνοι που εργάζονται στο Ίστμαν πρέπει να φύγουν από το κτίριο. Γιατί, για να το πω προσεκτικά, κοντεύει να τους πλακώσει το κτίριο υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι να μεταφερθούν σε άλλο κτίριο. Γιατί είναι και δύσκολες συνθήκες κατά τις οποίες δουλεύουν. Το κτίριο Eastman λοιπόν στεγάζει μέχρι σήμερα το διαμεσολαβητή, το ελεκτικό συνέδριο και τον επόπτη προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων. Η μισή είναι στο Ίσπαν και η μισή είναι στο Μοντουαγέ 63. Ε, το μισθωτήριο συμβόλαιο για το Μοντουαγέ 63 λύγει ε, στα τέλη του 2012. Ελέγχεται τώρα το ενδεχόμενο μπορεί να παραταθεί για μικρό χρονικό διάστημα, έτσι και αλλιώς πρέπει να φύγουν κάποτε. Η τιμή που πληρώνουμε σήμερα είναι 191 ευρώ το τετραγωνικό επειδή ο διαμεσολαβητής στο ελεγκτικό συνέδριο και ο πόπτης προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν έχουν επομιστεί το πλήρες κόστος που θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε ως μίσθωμα. Εντάξει, πληρώνουν τα κοινόχρηστα, που πούμε, το ε, ρεύμα, τη θέρμανση ε, και δεν θα είναι όλα ουδέτερα για τον προπολογισμό. Και υπάρχει μια προσημείωση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που οδηγεί σε μεγάλες παρανοήσεις και στο μέλλον και ο διαμεσολαβητής αλλά και ο υπόπτης δεδομένων καθώς επίσης και το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να επομίζονται το κόστος που δημιουργούν οι ίδιοι για τις δικές τους δραστηριότητες. Λοιπόν, και κάπως καθαρίζει και αυτή η φαιά ζώνη που ισχύει αυτό τον καιρό στο κτίριο Eastman. Πώς έχει τώρα η κατάσταση? Έχει γίνει πλέον αφόρητη, το γνωρίζουμε. Το εμβαδό είναι 5.789 ε, τετραγωνικά, ε, στο Μοντουαγέ είναι 7.506 τετραγωνικά. Το κόστος για το Σιάνς Μοντουαγέ, το κτίριο, είναι ετήσιος 1.166.144 με τιμα αριθμική αναπροσαρμογή και το ποσοστό που αναλογεί στο εκάστοτε όργανο θα το επομίζονται και οι ενδιαφερόμενοι, οπότε δεν θα έχει επιπλέον κόστος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μόνο που πληρώνουμε εμείς είναι το κόστος ασφαλείας, γιατί έτσι κι αλλιώς ε, θα το πληρώναμε αν έχουμε δικούς μας υπαλλήλου σε αυτά τα κτίρια. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, συνεισηγητέ και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε τώρα να σα διαβάζω αριθμού, γιατί ο καθένα μπορεί να τι βρει στο διαδίκτυο σε λεπτομέρειε. Γενικώ πάντω, για μας Το πρώτο αρχικό κόστος θα είναι 2 εκατομμύρια 200 περίπου και ε, θα έχουμε ένα συμβόλαιο για 21 ε, έτη, έχουν γνωμοδοτήσει και εμπειρογνώμονες. Βέβαια αυτές οι γνωματεύσεις δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες, είναι λίγο συγκεκριμένες, να το πούμε στη διοίκηση. Γιατί λέω ότι δεν είναι τόσο καθαρές, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς αυτό θα επηρεάσει το ρετήσιο προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Τα έχουμε υπολογίσει όλα αυτά με τρόπο πάρα πολύ περίπλοκο, αλλά το κόστος που αναφέρεται εκεί πιστεύουμε ότι έχει υπολογιστεί σωστά. Δεν θα σας πω όλες αυτές τις περίπλοκες εμ, ε, εξισώσεις και τους προϋπολογισμούς. Ε, μπήκε σε αυτό τον κόπο και τη βάσανο η δική μου συνεργάτης. Ε, πάντως θεωρούμε ότι είναι λογικά αυτά που προτείνονται και στο μέλλον 5.300 τετραγωνικά ε, θα έχουμε ε, ε, υπέργεια επιφάνεια και 1.500 υπόγεια και οι υπάλληλοι δικοί μας θα είναι σε κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε κτίρια που ήδη έχουμε μισθώσει ή έχουμε ήδη αγοράσει. Τιμό λέγεται ο ιδιοκτήτης, ε, έχει χτιστεί το κτίριο στις αρχές δεκαετίας του 60, αλλά κενίστηκε πλήρως. Ε, έχει ε, γίνει κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης και μελέτη για το έδαφος, για τη, τα πατώματα, τη ρήπανση. Βρέθηκε αμίαντος, αφαιρέθηκε ε, και υπάρχει πιστοποιητικό ελεύθερο αμοιάντου, Asbestos safe, οπότε δεν θα χρειαστεί εδώ να γνωμοδοτήσουμε γιατί θεωρώ ότι έχουν γίνει όλα σωστά και επιτέλους ε, ο διαμεσολαβητής και τα άλλα θεσμικά όργανα θα πρέπει να βγουν από το Eastman και να μετακομίσουν κάπου οι υπηρεσίες αυτές. Νομίζω ότι από πλευρά τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει γίνει καλή δουλειά για αυτά τα κτίρια. Ευχαριστούμε κυρία εισηγήτρια. Ποιος άλλος για το ίδιο θέμα. Το κτίριο Σιάνς Μοντουαγέ. Προτείνω να μην γνωμοδοτήσουμε. Ο Γιώργος Λάιον. Ένα ερώτημα, δεν διαφωνώ. Το Μοντουαγέ είπαμε. Ξέρετε ότι το ελεγκτικό συνέδριο, ο διαμεσολαβητής, χρησιμοποιεί τον χώρο αυτό, αλλά τι κόστος θα είχε η απομάκρυνση του για το Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχει εδώ συνδιαχείριση. Merci. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question de notre vice-président Μπορεί να απαντήσει κάποιο στην ερώτηση αυτή του αντιπρόεδρου, η συγκήτριά μα που σε όλα απαντά. Έχω φέρει τα έγγραφα. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 22,78%. Δεν έχω τα ακριβή ποσά τώρα ε, αναλύσει. Τα έχω όμως για το συνολικό κόστος είναι 1.166.000. Οπότε υπολογίζεται το 22,78% για το μίσθωμα και τις λειτουργικές δαπάνες ε, είναι 80.541 ευρώ και συνολικά 346 και κάτι ψηλά. Για τον επόπτη 86.000 Ενεκτικό συνέδριο 63.000 και 314 341 συγγνώμη, χιλιάδες ο διαμεσολαβητής. Ε, η Γενική Διεύθυνση εκπροσωπείται εδώ. Μπορεί κάποιος να μας δώσει ε, τα στοιχεία που ρώτησε και ζήτησε ο κύριος Λάιον συμπληρωματικά στα όσα μας είπε η συγκήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αριθμοί που ανέφερε η συγγήθρια είναι ε, προφανώς σωστή. 22% περίπου αναλογούν στο κοινοβούλιο του εμβαδού, έτσι. Είναι περίπου 350.000 ευρώ. 35 ε, με 40 υπάλληλοι εγκαθίστανται εκεί έτσι και έτσι έχουμε πρόβλημα έλλειψη γραφείων στις Βρυξέλλες και χαιρόμαστε που μπορούμε να ε, εγκαταστήσουμε εκεί 35 με 40 υπαλλήλους του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, από εκεί και πέρα τι κάνουμε. Η συγγήτρια προτείνει να μην γνωμοδοτήσουμε για το κτίριο Σιάνσμα του ΑΓΕ. Εντάξει, καλώς. Εντάξει. Στη συνεδρίασή μας στις 31ης θα εξετάσουμε ο συνήθως μια γραπτή διγνωμοδότηση για το σχέδιο διευθέτησης του κτηρίου Eastman, το Eastman Building που λέμε. Λοιπόν, σας προτείνω τώρα να σταματήσουμε για δύο λεπτά μέχρι να έρθει ο πρόεδρος Τόιρερ. Ο κύριος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 Du brauchst sie nicht. See you. Voilà, mes chers collègues, je remercie le président. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον πρόεδρο Τόιρερ που προσήλθε. Η συνεδρίασή μας τώρα είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Μαζί με τους συντονιστές θελήσαμε να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων ως προς το δημοσιονομικό κανονισμό. Αύριο προβλέπεται να αρχίσει ξανά τριμερής διάλογος και καλό είναι να ξέρουμε πού βρισκόμαστε ώστε και οι δύο μας επιτροπές να τα γνωρίζουν αν θέλετε κι εσείς να θέσετε ερωτήματα κτλ. Η Ινγκε έχει το λόγο. Με ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια μας κάνει εντύπωση ότι η πρόεδρη ε, ε, δεν είναι. Κυρία Ιβάνοβα, χαίρομαι που ασχολείται με αυτά τα θέματα, γιατί οι γυναίκες έχουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση στον προπολογισμό. Οπότε αύριο ε, θα έχουμε ιδιαίτερη χαρά να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ε, θα χάσετε μια μεγάλη εκδήλωση. Κρίμα που οι πρόεδροι και οι άνδρες θα λείπουν. 14 είναι τα εκκρεμή ακόμα σημεία με διαφορετική στάθμιση και διαφορετικό μέγεθος. Υπάρχει ολόκληρο άρθρο δηλαδή όπου διαφωνούμε πάρα πολύ. Ας πούμε στη συνδιαχείριση το άρθρο 56, αλλά είναι και μια υποπαράγραφος ή υποπρόταση, ενώ σε άλλα σημεία ε, ε, που θα έχει το Συμβούλιο τον τελικό λόγο και τον καθοριστικό. Ως Κοινοβούλιο προχωρήσαμε αρκετά ε, και παραμένει καλή η ατμόσφαιρα εργασίας και θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να σταματήσουμε ε, τις χαρές και τις αγκαλιές και αύριο θα αρχίσουν τα ζόρια, για να το πω ναι. έτσι, ε, για την απαλλαγή. Το Κοινοβούλιο έχει με βάση τη συνθήκη το καθήκον να ασχοληθεί με την απαλλαγή και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το γράφουμε στον κανονισμό, το δημοσιονομικό. Έχουμε τροπολογίες να διαπραγματευτούμε του Συμβουλίου που το Συμβούλιο δεν κινείται καθόλου. Μέχρι τώρα λέμε ότι δίνουμε απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ε, ε, έχουμε εργαστεί και για τους άλλους οργανισμούς και τους άλλους φορείς. Αυτό δεν θέλει να το δεχτεί το Συμβούλιο και σημαίνει ότι θα πρέπει ε, όλα αυτά να ενταχθούν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για όνομα του Θεού, ας γίνει, εν περιπτώσει, αλλά θα έχει μεγάλο πρόβλημα η συζήτηση και η αντιπαράθεση και και το θέμα της πρόσβασής μας ε, στις εκθέσεις του εσωτερικού αναθεωρητή ε, της, ε, του κάθε έχουμε μια τροπολογία που λέει ότι μπορούμε να έχουμε υποπροϋποθέσεις πρόσβαση σε απόρριτα έγγραφα. Το Συμβούλιο αυτό το αφισβητεί. Παρόλο που με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ήδη συμφωνήσει η διαδικασία και θυμίζω ότι υπάρχει μια υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπου κάποιοι κανονικοί πολίτες έχουν ε, κερδίσει το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα και εφόσον το έχει ε, κερδίσει αυτός ένας πολίτης, πώς μπορεί κάποιος να αρνείται το δικαίωμα σε βουλευτές. Ε, και από εκεί πέρα δεν υπάρχει περιορισμός. Εμείς έχουμε βάλει περιορισμούς και όρους και προϋποθέσεις και θα χαθούν. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδε ότι είναι καλύτερο ε, να ακολουθεί τις δικές μας τροπολογίες παρά να σένεται στα δικαστήρια. Αλλά το Συμβούλιο όπως Σοφία νομίζω χωράει ακόμα βελτίωση. Άλλο θέμα στο οποίο θα διαπληκτιστούμε. Είναι θέματα δικής μας αρμοδιότητας Επιτροπής Προϋπολογισμών. Τι γίνεται με το υπόλοιπο προσεκαθάριση του προϋπολογισμού στο τέλος του έτους. Έχουμε τροπολογίες που λέμε ότι θέλουμε να μεταφέρονται αυτά στο επόμενο έτος Εκεί να δείτε τι θα γίνει <laughs> το Συμβούλιο. Τέταρτον, η εγγραφή στο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Έχουμε δύο τροπολογίες εκεί και συνεχίζουμε τον αγώνα. Στη συνέχεια, πέμπτο θέμα. Ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό εδώ στην Επιτροπή, τι γίνεται με τους εκτάκτους προϋπολογισμούς. Ας πούμε, αν δεν συμφωνήσουμε στη διαδικασία του προπολογισμού, έχουμε συμβαστική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι με 12 τιμόρια μπορεί να λειτουργεί εκτάκτο ο προπολογισμό μόνο για τέσσερι μήνε. και μετά να υποχρεούται το Συμβούλιο να έρχεται και να το συζητάει. Το πρόβλημα είναι ότι στο μεταξύ μπορεί να έχουμε αντιευρωπαϊκέ κυβερνήσει, οι οποίες βρουν τα χέρια του και λένε δεν θέλουμε κοινοτικό προπολογισμό, κάντε 12 τιμόρια. Αυτό είναι μια πρόβλεψη για τη χειρότερη δυνατή περίπτωση και είναι πάρα πολύ ε, ε, λογικό και σόφρο να το ρυθμίσουμε σε περίπτωση που προκύψει κάτι τέτοιο. Άλλα θέματα που έχουμε στο πλευρό μας και σε αυτό το θέμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε τι θα βγάλει. Άρθρο 18, επίσης πολύ ωραίο. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τα πρόστιμα. Και... Δηλαδή, ή και θελοντικές πληρωμές, ας πούμε συμφωνίες για τον προϋπολογισμό, για τον καπνό έχουν πληρώσει με θελοντικέ ρυθμίσει καπνοβιομηχανίε. Και είπαμε να μπαίνει αυτό στον προπολογισμό τη Ένωση. Το Συμβούλιο ούτε να τα ακούσει. No go. Άλλο θέμα. Έβδομο. Εκεί γίνονται πιο άνετα τα πράγματα, μεταφορέ πιστώσεων και έχουμε κάνει τροπολογίε που μειώνουν το, τη γραφειοκρατία των μεταφορών πιστώσεων, αλλά το θέμα τι γίνεται με τις δύο τελευταίες εβδομάδες του χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ε, ότι στα διαρθρωτικά ταμεία είναι πολλές οι πληρωμές, αλλά δεν μπορούν να γίνουν ε, μεταφορές πιστώσεων γιατί δεν συνεδριάζει πια η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Και μας λένε, δώστε μας μια γενική εξουσιοδότηση, ένα εξούσιο ε, το τελευταίο δεκαεπενθήμερο κάθε έτους, να κάνουμε ό,τι θέλουμε τα κονδύλια. Δεν θέλουμε να το κάνουμε εμεί αυτό, ούτε το Συμβούλιο. Και προτείναμε να δημιουργήσουμε ένα 13ο μήνα, όπου το Γενάρη να μπορούμε να κάνουμε από το προηγούμενο έτος τη μεταφορά πιστώσεων, να διατηρείται ο ενιάυσιος προηγουμενο ετος τη μεταφορα πιστωσεων να διατηρειται ο ενιαψιο χαρακτήρα του προπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα βρίσκει ε, περίεργα. Θα τα πει το Συμβούλιο. Το θέμα είναι αν θα δημιουργήσουμε ενα 13ο μήνα ή όχι, αν δεν θέλουν αυτό να μα πούν τι θέλουν. Άρθρο 30 το αγαπημένο μου άρθρο, το έχω τονίσει. Ποιος επιτρέπεται να υπογράψει τον προπολογισμό όταν έχει ολοκληρωθεί. Η συνθήκη λέει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ κάθισα ώρες ολόκληρες και άκουσα το κήρυγμα ε, ε, της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου που να μου λένε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συνθήκη με δημοσιονομικό κανονισμό έρχεται και το προτείνει το Συμβούλιο αυτό. Τι προτείνει. Ότι Κάποιο πρέπει να υπογράφει το προπολογισμό. Δεν λέει ο πρόεδρο του κοινοβουλίου ποιο να είναι. Και πάλι υπάρχει προσφυγή του Συμβουλίου στο δικαστήριο που εκκρεμεί. Πολύ δύσκολο. Δύο πράγματα που πρέπει να πω που μου δημιουργούν περίεργα αντανακλαστικά και γελάω κάθε φορά. Και αυτό θα το συζητήσουμε. Τώρα σοβαρεύουν τα πράγματα στο άρθρο 131, το χρηματοδοτικό μέσο και το θέμα αν μπορούν τα χρηματοδοτικά μέσα να ε, κάνουν revolving, δηλαδή να επαναχρησιμοποιούνται. Αλλιώς ε, δεν έχει νόημα το χρηματοδοτικό μέσο. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο κείμενο και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καλό το κείμενο. Αλλά φροντίσαμε η Επιτροπή Προπολογισμών και οι επιμέρου επιτροπέ να έχουν όσο γίνεται περισσότερο λόγο για το ύψο του ποσού που χρησιμοποιείται. Κάθε χρόνο στον προπολογισμό το αποφασίζουμε από την αρχή. Υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα που είναι, πηγαίνουν καλά και άλλα που δεν λειτουργούν τόσο καλά. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα κάθε χρόνο να ορίζουμε τα ποσά στις γραμμές του προπολογισμού. Δηλαδή, να υπάρχει μια μέγιστη δυνατή διαφάνεια και δυνατότητα ε, συμμετοχής της δημοσιονομικής αρχής. Και τα δύο αυτά είναι καλά μέτρα, έτσι ώστε και για αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα να μπορέσουμε να δώσουμε μια καλή και θετική άποψη. Βρήκαμε καλές λύσεις και διαπραγματευτήκαμε. Κάτι άλλο που παραμένει σε εκκρεμότητα, το άρθρο 178, Trust Funds, μεγάλο εργοτάξιο, λατομείο ολόκληρο είναι. Ε, το Συμβούλιο προσπαθεί εκεί να ε, προχωρήσει πάρα πολύ περιοριστικά. Εγώ δεν έχω ξαναδεί νομικό κείμενο που να αρχίζει με τη λέξη «απαγορεύεται». Έτσι αρχίζει. Ε, έτσι λέει το Συμβούλιο. Απαγορεύεται το εξή, το τάδε και το δίνα. Εδώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πολλή δουλειά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει trust όχι μόνο ανθρωπιστικά, αλλά και θεματικές δράσεις, ας κλιματική αλλαγή και τέτοια. το Συμβούλιο έχει φτιάξει ένα κείμενο που λέει ότι εφαρμοστικέ ε, αρμοδιότητε έχει μόνο το Συμβούλιο, τέλεια, εκτελεστικέ. Δεν είναι αυτό η αγαπημένη διατύπωση για τους βουλευτέ. Άρθρο 195 τα κτίρια. Δεν ξέρω αν η Ένωση μπορεί να συνάπτει δάνεια μόνο για τα κτίρια. Καλό θα ήταν να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα, θα ήταν πιο φθηνά τα πράγματα. Και το Συμβούλιο νομίζω αύριο πρέπει να αναθεωρήσει λίγο τη θέση του. Και εκεί βάλαμε πολύ περισσότερη διαφάνεια και χάρη στην εισηγήτριά μας για τα ακίνητα στο θέμα της συναπόφασης και όχι συναπόφασης, δηλαδή να έχει λόγο η Επιτροπή Προϋπολογισμών και από νωρίς. Και το θέμα είναι τώρα τα κατώτατα όρια, από, από ποιο ε, ποσό και μετά. Δεν έχει καταλήξει ακόμα αυτή η προσπάθεια. Κάτι άλλο που εκκρεμεί όχι για αύριο, αλλά για αργότερα, το άρθρο 156, η συνδιαχείριση των πόρων, και αυτό είναι μεγάλο εργοτάξιο, δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά αν ο καθένας κινηθεί προς την κατεύθυνση του άλλου δεν είναι ανυπέρβλητα τα εμπόδια. Αλλά επειδή είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα, ε, είναι ε, τι δικαίωμα ελέγχου έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι υποχρεώσεις ελέγχου έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και έχουμε και πολιτικούς στόχους με αυτό το share management. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι και στην Ελλάδα και στην Ισπανία πολύ περισσότερο το βλέπουμε από όσο θα θέλαμε να το βλέπουμε. Στο άρθρο 117α, επιδοτήσεις και τι γίνεται με το ΦΠΑ. Εμείς θέλουμε στο μέλλον το ΦΠΑ να μην επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είναι η άμεση, αυτό θα ισχύει μόνο για την άμεση διαχείριση, όχι για τη συνδιαχείριση, δηλαδή μόνο για την έρευνα. Δηλαδή, εκεί που επιδοτούμε κάποια προγράμματα ή κάποια έργα να μην ε, επιβάλλεται φόρος θέμενη αξίας. Και το τελευταίο κατά τη πράξης και αυτό εκκρεμεί και μέχρι τελευταία στιγμή θα εκκρεμεί. Μέχρι τώρα υπάρχει μια διοικητική συμφωνία, common understanding, αλλά δεν λύνει το ερώτημα ότι τι θα κάνουμε αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για ε, τις κατεξουδότηση πράξη. Αλλά η δημοσιονομική αρχή χρειάζεται πράξεις εξουσιοδότηση. Είναι πραγματικά το φιλί της ζωής. Στην πολιτική έχω ζήσει την εξή εμπειρία. Όταν συνεννοούμαστε καλά μεταξύ μας δεν χρειάζονται κανόνες. Οι κανόνες είναι για τη χειρότερη δυνατή περίπτωση και γι' αυτό θα πρέπει να θεσπιστούν πολλοί διαφωνούν με αυτά που προτείνουμε, δεν πειράζει. Καμιά φορά χρειάζεται χρόνος για να πιστούν. Έτσι έχουν τα πράγματα, θα μπορούσαν να έχουν και πολύ χειρότερα. Προγραμματισμός τώρα, χρονοδιάγραμμα αύριο, ε, τριμερής διάλογος και την 1η Ιουνίου και ενδεχομένως 12 Ιουνίου στο Στρασβούργο υπάρχει και αυτή η ημερομηνία χρειαστή. Κατά τα άλλα, χτες ως εισηγήτρια συναντήθηκα ε, με την Όλαφ στο τριμερή Λογώ και δεν βλέπω μόνο ε, φως στην άκρη του τούνελ, αλλά ο ήλιος λάμπει, δηλαδή είναι κοντά το τέλος και σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Βλέπω εδώ τους διπλανούς μου να οδοκροτούν θορυβοδός. Μένουν ακόμη 14 θέματα βέβαια και σημεία και επί των περισσότερων υπάρχει κοινό μέτωπο Κομισιόν Κοινοβουλίου και οι δυσκολίε έγκυνται στο Συμβούλιο. Κυρία Μπραντνερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ σύντομα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ ε, για τις διαπραγματεύσεις και τη διαπραγματευτική τέχνη της ε, εισηγήτριας και τη στρατηγική της ακριβώς αυτό το θέμα της διαχείρισης ε, θα πρέπει να έχουμε προτεραιότητες και για τα external trust funds, το συζητήσαμε και το πρωί, το θεωρώ παράλογο στην εξωτερική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, χρηματοδοτεί τόσα τέτοια καταπιστεύματα της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΗΕ και εμείς φωνάζουμε στην Επιτροπή Ελέγχου ότι δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν τα κονδύλια, ότι δεν έχουμε καμία ορατότητα η Κομισιόν λέει, ωραία, να φτιάξουμε δικό μας trust fund, να το διαχειρίζετε και να έχετε εσείς περισσότερο έλεγχο και ορατότητα. Και τώρα έρχονται τα κράτη-μέλη και λένε, αποκλείεται. Ε, κάπου, τι θα γίνει τώρα. Ε, είναι το θέατρο του παραλόγου. Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Αν δεν το θέλουν, τότε να σταματήσουμε να το επικρίνουν. Αυτό που κάνει τα χρήματα Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή. Γιατί Καμιά φορά έχει νόημα να συνεργάζεται κανεί και να φτιάχνει τέτοια ταμεία, όχι μόνο για έκτακτε ανάγκε, αλλά α πούμε για την ελονοσία, το AIDS, ε, συνεργασία με τον ΟΗΕ. Γίνεται μεγάλη κριτική που πηγαίνουν τα λεφτά. Και τώρα που η Κομισιόν λέει θα φτιάξει το δικό μου μέσο, γρινιάζουν τα κράτη-μέλη και το απορρίπτουν από χέρι. Καμιά φορά με εκπλήσουν όλα αυτά τα πράγματα ναι. διαμαρτύρονται συνεχώς και γκρινιάζουν ε, οι αρμόδιοι της ε, ε, εξωτερικής πολιτικής, αλλά όταν πρόκειται για τους ειδικού για τα οικονομικά αντιδρούν. Και έρχεται κάθε Προεδρία του Συμβουλίου και διαμαρτύρεται σε εμά. Θα πρέπει να διαμαρτύρεται στα Υπουργεία της. Ένα μικρό σημείο, δεν ήταν στις 14, ε, και αυτό που είπε η κυρία Νέτσχη προηγουμένως, πώς ορίζεται η κρίση ή η επίγουσα κατάσταση. Ως κοινοβούλιο ε, κάναμε μια πρόταση, βέβαια θα το λύσει ο δημοσιομικός κανονισμός αυτό για να έχουμε μια πιο ενιαία θέση. Και ε, αν το κατάλαβα καλά, και πάλι αυτό κατέληξε στις εξουσιοδότηση πράξης, που έχει το εξή κίνδυνο. Να μην μπορεί να ρυθμιστεί ενιαία από τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το βγάλουμε το είπε και η κυρία Νέτσχη προηγουμένως, να έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση γενικότερη. Ξέρω ότι αυτό δεν θα συζητηθεί αύριο, αλλά επειδή το συζητήσαμε προηγουμένως, ήθελα να το θέσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα... Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμασού, Καταρχά, σα ευχαριστώ πολύ και την κυρία Γκρέσλα, η της Επιτροπής Προπολογισμών. Ο συνάδελφος Ριβελίνη επίσης ε, συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση θα ήθελα να πω ότι μπορεί να είναι αποφασιστικό αυτό το σημείο γιατί ε, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κονδύλια ε, στο μέλλον που να διαφεύγουν του ελέγχου μας ε, και με τα σφάλματα που έχουν ε, προκύψει θα πρέπει οπωσδήποτε να τα ελέγχουμε. Το είδαμε και στην Επιτροπή Ελέγχου Προπλογισμού. Ξέρω την Ίγκε Κρέσλε και είμαι βέβαιος ότι ε, έχει ιεραρχήσει σωστά τα θέματα. Δυστυχώς που θα λείπω αύριο. Το πρωί θα μπορούσα. Έχω σημαίνει στην 1η Ιουνίου θα έρθω οπωσδήποτε. Αλλά και ως κοινοβούλιο γενικά θα πρέπει να συνταχθούμε και να ε, προχωρήσουμε από κοινού. Και να αποφασίσει και Ολομέλεια. Και μπορεί και παραπίδα να υποκύψει στη γοητεία της διαπραγμάτευσης ε, το Συμβούλιο και να συμφωνήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει κάποιος μη Γερμανός ο οποίος θα ήθελε το λόγο. Παρατηρώ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έχω κάθε θαυμασμό προς τους Γερμανούς συναδέλφους, παρακολουθά με τρομερή προσοχή. Εφόσον λοιπόν δεν ζητάει το λόγο κάποιος άλλος, θα κάνω μία παρατήρηση και θα θέσω μία ερώτηση στην εισηγήτρια. Η παρατήρηση είναι ότι Παρακολούθησα με προσοχή τα 14 θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα και τουλάχιστον δύο από αυτά, αν πρόσεξα καλά, είναι θέματα που άπτονται του δημοσιονομικού κανονισμού και τα οποία θα αναφερθούν και στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό. Πρόκειται για τα υπόλοιπα τα δημοσιονομικά είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αιτήσια βάση μετά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και κάθε χρόνο έχουμε πολλούς, δισ ε, πολλούς δισταγμούς για τον τελευταίο διορθωτικό που στην ουσία παραπέμπει, ξαναστέλνει στους 27 υπουργούς τα πλεονάσματα τα οποία η καλή διαχείριση ή η κακή διαχείριση, διότι δεν μπόρεσαν να τα χρησιμοποιήσουν σωστά, επέτρεψε να εξοικονομηθούν σαν ποσά. Αυτά τα υπόλοιπα λοιπόν σε αιτήσια βάση είναι ένα μείζον πρόβλημα, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση που έχουμε προβλήματα για τη χρηματοδότηση των νέων πολιτικών. Ταυτόχρονα αναφερθήκατε στην δημοσιονομική χρήση εισαγωγικά των νέων ταμείων, πάνω στο οποίο θέμα θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του MFF. Πρόκειται για ένα κοινό στόχο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, φλέγεται λιγότερο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επαναντάξει το Ταμείο Ανάπτυξης στον κοινό προϋπολογισμό και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να δημιουργηθούν δορυφορικοί προϋπολογισμοί εν πωλής, διαφεύγοντας του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ορισμένα προγράμματα όπως το ΙΤΑ ή το GMS. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε αυτές τις τακτικές συναντήσεις για να συντονίζουμε καλύτερα τις θέσεις που ε, έχουμε στα πλαίσια των παραλλήλων διαπραγματεύσεων. Αυτή ήταν η παρατήρηση. Η ερώτηση αφορά το χρονοδιάγραμμα. Παρατήρησε αυτά που είπατε αύριο την 1η Ιουνίου, ο επόμενος τριμερής διάλογος, θα υπάρξει και η συνάντηση για την ΟΛΑΦ. Ποιες είναι οι προοπτικές που ανοίγονται χρονικά για να υπάρξει μία κάποια συμφωνία γιατί κάποια στιγμή θα τεθεί το θέμα εάν θα ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση και αν θα καταλήξουμε σε μια κανονική διαδικασία ή μήπως εάν πιστεύετε ότι μέσω της πλέον πραγματιστικής διαδικασίας και υπομονετικής που έχουμε ξεκινήσει θα καταλήξουμε μέσα σε ένα λογικό χρόνο τη διαπραγμάτευση. Για να απαντήσω στη Φρανσίσκα θα ήθελα να πω ότι η προσπάθεια καθορισμού της κρίσης ήταν κάτι το πάρα πολύ δύσκολο και θα το συζητήσω μαζί της και σε κάποια άλλη φάση. Πάντως δεν είχαμε πάρα πολλά εφικτά θα έλεγα μπροστά μας για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τους ενδιαφερομένους σχετικά με την εφαρμογή αυτού του τμήματος του κανονισμού. Ο κανονισμός αυτός ε, είναι, θα έλεγα πρέπει να εφαρμοστεί. Το 40% των υπαλλήλων της Επιτροπής εργάζονται με αυτό το κώδικα, οπότε πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ γενικόλογη και θολή θα έλεγα η διαδικασία και δεν μπορέσαμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εγώ προσπαθώ να υπάρξει μια κάποια συμφωνία. Χρειάστηκε πάρα πολλές χρόνος Προσπάθησαν πάρα πολύ όλοι, ευχαριστώ και τη Γραμματεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη δική μου Γραμματεία. Όλοι έκαναν τεράστιες προσπάθειες, εν για μια τέτοια συμφωνία. Είναι εφικτή. Πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό υλικό σε αυτήν τη φάση για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Πάντως υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες τι θα κάνουμε με τις τροφολογίες MFF αν το Συμβούλιο δεν τις δεχτεί. Μπορώ να τις μεταφέρω απλά στο Ράιμερ, ευχόμενοι απλά τύχη καλή, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Έχω επίσης την αίσθηση ότι οι αρχηγοί κρατών δεν μπορούν να συνεννοηθούν για το θέμα το αυτά με τα υπουργεία τους. Η δική μου χώρα, η κυρία Μέρκελ σαν παράδειγμα, πηγαίνει στη συνάντηση κορυφής και εκεί λέγεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται όλος ο κοινοτικό προϋπολογισμός για την ανάπτυξη. Μετά λέω ότι έκανα προτάσεις, αλλά το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας αρνείται τις προτάσεις αυτές. Αυτό επαληθεύεται πάρα πολύ συχνά πηγαίνω εκεί, έρχομαι σε επαφή μαζί τους, ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο και με κοίταγαν λίγο περίεργα. Υπάρχουν κάποια πράγματα λοιπόν τα οποία δεν κατανοώ εύκολα. Θεωρώ ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ στο τέλος του χρόνου. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί αλλιώς θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα, θα υπάρξει πολλαπλασιασμός κανόνων στα εξειδικευμένα ταμεία, ήδη έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με το 57, η ψηφοφορία έφτασε στην Περιφερειακή Επιτροπή και ε, η καθυστέρηση δεν είναι δικό μου λάθος. Το Συμβούλιο δυστυχώς μέχρι τώρα δεν στάθηκε ικανό να πάρει αδίποτε απόφαση σε σχέση με το 56 μάλλον. Ε, και κάθε φορά ζητάει να τεθεί σαν πρώτο θέμα σε συζήτηση την επόμενη φορά. Πρέπει λοιπόν να τεθεί σε ισχύ για να ξεκαθαρίσουν ορισμένα κάποια προβλήματα. Ε, για τα επιλέξιμα κόστη σαν παράδειγμα. Έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα πλέον και η διαχείριση των ταμείων θα βελτιωθεί αρκεί να υπάρξει ένας εξορθολογισμός των κανόνων σε όλα τα ταμεία και αρκεί να μην υπάρχουν αντιφάσεις. Και θα πρέπει επίσης να ερμηνευθούν οι κανόνες ανάλογα με τα ταμεία. Ο δημοσιονομικός κανονισμός, σαν παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθεί από το ελεγκτικό συνέδριο ενώ οι υπόλοιπε υπηρεσίε θα χρησιμοποιούν τους εξειδικευμένου κανονισμού. Κοιτάξτε, συντηρούμε στην ουσία μια τεράστια γραφειοκρατία λόγω ακριβώ των επιμέρου προγραμμάτων έρευνα. και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και η Προεδρία της Δανίας θέλει μια κάποια συμφωνία Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υπάρξει συμφωνία. Αλλά πάντως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να περάσουν. Και αυτό ίσως να πω και στους φίλους του Συμβουλίου που είναι παρόντες στις συναντήσεις μας, ενώ εμείς δεν είμαστε παρόντες στις δικές τους συναντήσεις, εμείς καταθέσαμε τις τοπολογίες αυτές και το λέω για το Συμβούλιο για να λύσουμε τα προβλήματα, γιατί από ό,τι φαίνεται είμαστε οι μόνοι που θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Γι' αυτό προσπαθούμε και γι' αυτό πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε επίπεδο λεπτομέρειας, γιατί ο προπολογισμό είναι λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, το θέμα να κλείσει γρήγορα. Σε ευχαριστώ, Ίγκε. Ε, μένουμε όλοι έκθαμβοι. Έχεις κάνει ε, τρομερή δουλειά και με ε, τη γραμματεία και με τους δύο συναδέλφους που παρακολουθούν τα θέματα αυτά πάρα πολύ. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Ραντεβού την Πέμπτη το απόγευμα. Τελευταία ενημέρωση. Οι φίλοι του Μιγγέλ Πόρτας, του εκλειπών του συναδέλφου μας διοργανώνω ένα μικρό μνημόσυνο, μια μικρή τελετή την Πέμπτη το πρωί στις 9, εδώ στο παρόν κτίριο, ε, στον πρώτο όροφο, στο χώρο Γεχούντι Μενουχή. Μισή ώρα. Αύριο, βεβαίως, κατά την έναρξη της Μήνης Συνόδου, ο πρόεδρος Σούλτς θα ε, τηρήσει ενός λεπτού σιγή και θα πει για δύο λόγια ε, προς μήν ε, του συναδέλφου που επιβίωσε. Είστε όλοι προσκεκλημένοι την Πέμπτη, αν θέλετε, συμμετάσχετε σε αυτή τη μικρή τελετή. Ευχαριστώ. Λήξη συνεδρίαση.